Καλησπέρα σας. Ας ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Σας καλωσορίζω όλους θερμά, βουλευτές και επισκέπτες, καθώς και όσους μας παρακολουθούν από το webstream, γιατί έχουμε την συνεδρίαση και με την παρουσία του κύριου Στόιβερ στο διαδίκτυο. Μια σειρά από ψηφοφορίες μας περιμένει. Έχουμε να συστήσουμε και μια γνωμοδότηση, αλλά πρώτα με μεγάλη χαρά καλωσορίζω θερμά τον δόκτωρα Στόιμπερ με μια μεγάλη και δικαιοκριμένη ε, πολιτική αεροδρομία πάνω απ' όλα ως Πρωθυπουργός του κρατήριου της Βαβαρίας αλλά και από το 2007 ως επικεφαλής της ομάδας ε, του υψηλού επίπεδου γιατί ο διοικητικό άχθος έχει ξαναέρθει στην Επιτροπή μας να μιλήσει στις αρχές αυτής της θητείας. Έχει παρακολουθήσει, όπως ξέρετε, πολύ καλά προσεκτικά την ποιότητα της δουλειάς μας και θα είναι, φαντάζομαι, και στην ομάδα που θα διατυπώσει ε, τον αντίκτυπο επιπτώσεων του έργου αυτού. Έχουμε πολλές νομοθετικές προτάσεις λοιπόν που χρειάζονται αξιολόγηση αντικτύπου και σήμερα το απόγευμα επίσης. Αλλά και δουλειά προπαρασκευαστική των νομοθετημάτων όπου προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εξέταση των συνεπειών προκατακτικά και να ενισχύσουμε την νομοθετική μας ε, αρμοδιότητα. και να βελτιώσουμε τις νομοθετικές μας ε, προτάσεις. Η τελευταία πρόταση για τις ε, δημόσιες προμήθειες ήταν νομίζω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει μια πρώτη ανάγνωση διεξοδικά, δώσαμε αρκετό χρόνο, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να αφήσουμε και να καθυστερήσει η διαδικασία. Ελπίζω να σας ενδιαφέρουν όλους το ίδιο αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε εδώ κύριε Στόιμπερ και θα έχουν βέβαια και οι συνάδελφοι την ευκαιρία να δείτε πόσο τις ερωτήσεις τους με τη σειρά. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Χάρμπορ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, χαίρομαι που έχω και πάλι την ευκαιρία, γιατί νομίζω ότι στην Επιτροπή σας είχα έρθει πριν από τέσσερα χρόνια. Χαίρομαι λοιπόν που έχω την ευκαιρία να μιλήσω μέσα για το θέμα αυτό του διοικητικού φόρτου Μετά από δύο χρόνια διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Μπαρόσο, πέρασαν συνολικά 7 χρόνια. Συνεχίζεται φυσικά αυτή η δουλειά, ανεξάντλητο το θέμα και ίσως να μην είναι και η τελευταία φορά που θα είμαι εδώ παρόν. Το θέμα, όσο κι αν εγώ ίσως να μην έρθω, θα σας απασχολήσει και θα περάσω μέσω συνμέντια και να πω γιατί πρέπει κανείς να αναλάβει ως επίτιμος εκπρόσωπος το θέμα αυτό. Έχουμε τουλάχιστον τέσσερι φορέ, έχω εγώ τουλάχιστον τέσσερι φορέ την εβδομάδα το καθήκον να ασχοληθώ με τα θέματα αυτά. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί και το λέω και το επαναλαμβάνω, διότι συμφωνούμε ότι η καθοριστική πτυχή για την αποδιάρθρωση αυτού του διοικητικού φόρτου είναι η πολιτική διάσταση η οποία βεβαίως έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις σήμερα. Και αν δούμε και αυτά που λέει ο Πρόεδρος, διαπιστώνουμε ότι ε, μεγάλοι επίτροποι που ενώπιον του Κοινοβουλίου καλούν ε, για περιορισμό της γραφειοκρατίας, επί παραδείγματι ομιλία του συνάδελφου Μπαρνιέ από το Δουβλίνο, όπου είχε προσέλθει ως υποψήφιος, υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πρέπει να πω ότι με ε, συγκίνησε πολύ ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε ο κ. Μπαρνιέ να καταγράψει τα σημεία στα οποία χρειάζεται να περιοριστεί η γραφειοκρατία, αλλά βέβαια και ο πρόεδρος Σούλτς, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει η Ευρώπη αντί να στέκεται πάνω στο κεφάλι, να στέκεται στα πόδια, και να μην ρυθμίζουμε πια τα πράγματα όπως τα ρυθμίζαμε παλιά, έχουμε κάνει σφάλματα κτλ. Και όλοι ρεν, με μεγάλη μου χαρά λέει ότι, γιατί και εκείνο απευθυνόμενο του Κοινοβούλου λέει ότι πάντοτε αγωνιζόταν για την, κατα... για την αποδιάρθρωση της γραφειοκρατίας θα κάνει ακόμη περισσότερα. Ο Γκίντερ Χιώτιγκερ, Γερμανός Επίτροπος, με την ίδια έμφαση και ούτω καθεξής. Τι θέλω να πω. Απερίφραστα ότι βεβαίως μπορεί αυτή η κατηγορία που απευθύνεται για την υπερβολική γραφειοκρατία να επηρεάζει την αποδεξιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαι λοιπόν επίτιμος πρόεδρος μεγάλου κόμματος στη Γερμανία και ως επίτιμος πρόεδρος είμαι περισσότερο παρατηρητής παρά παράγων της πολιτικής ζωής πλέον στη Γερμανία. Βλέποντας λοιπόν και δύο μήνες πριν από τις ευρωεκλογέ, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και το 1979 πρώτο πρώτο, την πρώτη χρονιά δηλαδή άμεσων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου πάντα βεβαίως εμφανίζονταν αντιευρωπαϊκά κόμματα, αλλά με πολύ περιορισμένη υποστήριξη από τους ψηφοφόρους, αυτή τη φορά βλέπουμε ότι μεγάλα ποσοστά αναμένεται να λάβουν τα κόμματα αυτά και δει στην Γαλλία με τη σειρά τα αναφέρω, μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε, μετά ε, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτω χώρε, σκανδιναβικά κράτη, αλλά και αν κοιτάξουμε και τις μαζικές εκδηλώσεις του Πέπε Κρίλο στην ε, Ιταλία, βλέπουμε ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στην Ευρώπη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, εάν δούμε στις προσεχείς εκλογές ποσοστό από 20 έως 25% της εκατοίκη περισσότερο ακόμη για κόμματα τα οποία είναι εκβάθρων κατά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την καταπολεμούν, τότε νομίζω ότι έχουν μπροστά τους τα θεσμικά όργανα των Βρυξελών πολύ μεγάλες προκλήσεις. Και γι' αυτό η ε, αποδιάρθρωση της γραφειοκρατίας θα είναι ένα τεράστιο έργο για να συμβάλλουμε επικοδομητικά στην αποδοχή από τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο θέμα του ευρώ θα τα αφήσω προς το παρόν εκτός, αλλά θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν στα υπόλοιπα θέματα όλο και περισσότερες πιέσεις ρυθμιστικές από τις Βρυξέλλες και αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια αίτια αυτών των αρνητικών εξελίξεων. Ιδάλλως δεν θα έθεταν το θέμα αυτό της, ε, του περιορισμού του διοικητικού φόρτου οι επίτροποι στις ομιλίες του. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει αυτή η τάση και η τοποθέτηση και ελπίζω ότι θα υλοποιηθεί και στην πράξη. με το ευρωβαρόματρο το οποίο γνωρίζω το τελευταίο, το έχω μελετήσει πολύ καλά, βλέπω ότι έχουμε από τη Γερμανία 40% των ερωτηθέντων σε ανοιχτό ερώτημα για το τι θεωρούν ε, ότι είναι το χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τι συσχετίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία το τέρα τη γραφειοκρατίας, γραφειοκρατικό φόρτος και Και στι κάτω χώρε, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σκανδιναβικέ χώρε, είναι τα ποσοστά εξίσου υψηλά. Σε δε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είναι το 1 τέταρτο. ένα- στου τέσσερι πολίτε θεωρεί ότι η Ευρώπη κατά κύριο λόγο σημαίνει γραφειοκρατία. Σε σχέση με το 2010 έχουν αυξηθεί σημαντικά αυτές οι τιμές. Η δε δήλωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει γραφειοκρατία σε ποσοστό έως και 74% βρίσκει σύμφωνους τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν και παρά την αυξανόμενη σημασία της Ευρώπης ε, για την ε, νομοθεσία, για τη ρύθμιση δηλαδή των ζητημάτων, η πολιτική συζήτηση στα κράτη-μέλη συχνά λαμβάνει χώρα χωρίς δυστυχώς να έχει ανταπόκριση στους πολίτες. Συστούνται τα θέματα στις Βρυξέλλες χωρίς να τα παρακολουθούν οι πολίτες, χωρίς να τα ε, γνωρίζουν. Και έτσι δεν υπάρχει η αποδοχή για τις όλο και περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Ενώ έχουμε ευρωπαϊκές ρυθμίσεις στον χώρο του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων, που ρυθμίζει και αντικαθιστά στο χώρο της εσωτερικής αγοράς τις διαφορετικές διατάξεις που ισχύουν στα 28 κράτη-μέλη. Αυτό διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και προωθεί, προωθείται από αυτές διαρκώς. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η ρήτρα εσωτερικής αγοράς της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται όλο και πιο διασταλτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χρησιμοποιηθεί, ε, για να αξιοποιηθεί για νομοθετική παρέμβαση σε όλο και περισσότερους τομείς. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με την στάση των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μια, όπως είπα, διαμαρτύρονται εν γέννη και συλλήβδην για τη γραφειοκρατία. Από την άλλη, ζητούν όλο και νέες διατάξεις και ρυθμίσεις σε νέους τομείς πολιτικής. Και έτσι χιλιάδες βουλευτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασχολούνται διαρκώς με την βελτίωση των ε, ρυθμίσεων. Με νέε ρυθμίσει, ιδιαίτερα σε περιπτώσει φυσικών καταστροφών, όπου απευθύνονται διαρκώ εκκλήσει για καλύτερε ρυθμίσει, αλλά και σε θέματα όπω η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι θεωρείται και είναι όντω σωστό αυτό ότι δεν έχουν γίνει αρκετά, δεν έχουν ληφθεί επαρκεί αποφάσει, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι στην καθημερινή ζωή, στα ζητήματα του καθημερινού βίου, δεν χρειάζονται νέε διατάξει. Έτσι λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε το εξής, ότι το κύριο και μεγάλο πρόβλημα είναι το πεδίο εξισορρόπησης μεταξύ της ε, αυτόνομης ευθύνης και της ε, αυτόνομης ρύθμισης των ζητημάτων, αλλά και αφετέρου της ασφάλειας. Δεν έχει και η ασφάλεια πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το, αυτή η λεπτή ισορροπία και το να πούμε ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα έχουμε το θάρρος να μην προβούμε σε ρύθμιση, αλλά και να έχουμε το θάρρος να λάβουμε αποφάσεις και να ρυθμίσουμε κάτι το οποίο χρειάζεται ρύθμιση, είναι ακριβώς το ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να ε, ενσκύψουμε και πάνω απ' όλα να γίνει η ε, γενική φιλοσοφική συζήτηση, η ακαδημαϊκή συζήτηση. Έχουμε λοιπόν στην Ευρώπη με τα 28 κράτη, 10 κράτη με, που αντιμετωπίζουν σοβαρή ε, οικονομική στασιμότητα, 10 κράτη που έχουν ε, αντιμετωπίσει ύφεση και μόνο 8 τα οποία παρουσιάζουν ανάπτυξη. Η οικονομική κρίση λοιπόν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί αυτή να δώσει λύσεις. Χρειάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα που να, καλύ... να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Και έχουμε ενημερωθεί στην ομάδα υψηλού επίπεδου για ένα κράτος, μάλιστα πρόσφατα, το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα πάντα με τη γραφειοκρατία, αλλά έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της Κύπρου και έχουμε ζητήσει από τους υπευθύνους να έρθουν να μας ε, πούν τι συμβαίνει εκεί. Ο επικεφαλής λοιπόν του Κυπριακού προγράμματος μας είπε ότι πέρυσι το 22% της, ε, του γραφειοκρατικού φόρτου ...125 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή εξοικονομήθηκαν. Και έχουμε επίσης τον περιορισμό των, ε, της χρήσης των επιταγών για τις πληρωμές σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί ήταν πολύ εκτεταμένη η χρήση των επιταγών. Αυτά ακούσαμε για την Κύπρο. Στη δε ομάδα υψηλού επίπεδου, κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια τη πρωτη θητειας θητείας, 2008-2009, και αυτό είναι το αρχικό μας, η αρχική μας εντολή, κοιτάξαμε καταρχάς τα, πιο σημαντικά, τα 13 πιο σημαντικά κεφάλαια πολιτικής στα οποία χρειάζεται να ε, μειωθεί η γραφειοκρατία. Εξετάσαμε 72 νομοθετήματα που αντιστοιχούν στο 20% περίπου του συνολικού δικαιοικού πλέγματος και ταυτόχρονα προκαλούν 80% της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης λόγω της υποχρέωσης για ενημέρωση που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό σημαίνει 124 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό το οποίο δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βάση δε ε, χρησιμοποιεί ακριβώς αυτά τα 20 νομοθετήματα, τα 20% νομοθετήματα τα οποία επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με 124 δισεκατομμύρια ευρώ και ως εκ τούτου το 80% του γραφειοκρατικού φόρτου. Και εδώ διατυπώνει η ομάδα μας 300 συγκεκριμένε προτάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν ε, μέχρι τώρα ε, εισαγάγει μέτρα τα οποία μπορούν να ε, αποφορτήσουν κατά 32,9 δισεκατομμύρια ευρώ τις 23 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν ορίσει έναν στόχο των 25, του 25% για μείωση αυτής της επιβάρυνσης και μάλιστα τον έχουμε υπερβεί στην πράξη. Δεν χρειάζεται να σας δώσω στοιχεία για τις επιμέρους ε, διατάξεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι η αναγνώριση των ηλεκτρονικών ε, αποδείξεων για την φορολογία που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις ε, φόρτιση κατά 18,4 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει εφαρμοστεί στα περισσότερα κράτη-μέλη, θα αναφερθώ δεξοδικότερα μετά. Επίσης, για τις, μικρότερες, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις μικροεπιχειρήσεις όπως λέμε, υποχρέωση για τον ισολογισμό και τη δημοσίευση των στοιχείων σημαίνει, η κατάργησή της σημαίνει ότι ε, αποφορτίζονται κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ οι επιβαρύνσεις αυτές. Έχουμε από την περίοδο δε, ε, του 2010 έως το 2012, δηλαδή στη δεύτερη μας θητεία, για πρώτη φορά την ε, εφαρμογή του υφισταμένου, έχουμε εξετάσει για πρώτη φορά πολύ προσεκτικά την εφαρμογή του υφισταμένου ευρωπαϊκού δικαίου στην, ε, στα κράτη-μέλη και έχουμε καταρτήσει μια έκθεση υλοποίησης, την έχετε και στα πρακτικά, στα έγγραφά σας και βλέπουμε ότι ένα τρίτο των γραφειοκρατικών δαπανών, του γραφειοκρατικού κόστους στην Ευρώπη, έγκυται οφείλεται στο γεγονό ότι ήταν ανεπιτυχή και αναποτελεσματική η υλοποίηση τη νομοθεσία επί επίπεδο κρατών μελών. Αυτό δυστυχώ είναι πολύ λίγο γνωστό. Και σε αυτό δυστυχώ η Ευρώπη δεν ασχολείται και επικρίνεται βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα προβλήματα, αλλά κατά βάση αυτό οφείλεται στην ε, στάση κρατών μελών όπως η Γερμανία και πολλά άλλα. Και έχω και κάποια παραδείγματα να προσφέρω. Επί παραδείγματι οι δημόσιες συμβάσεις μπορεί να κρατήσουν μέχρι 77 μέρες οι διαδικασίες του στη Λιθουανία και 241 ημέρες στη Μάλτα για να ολοκληρωθούν. Εάν λοιπόν τα κράτη-μέλη κατευθύνονταν προς την καλύτερη ε, δυνατή υλοποίηση, δηλαδή τις βέλτιστες πρακτικές όπως λέμε, της νομοθεσίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρούσαν αυτές τις προδιαγραφές, θα εξοικονομούσαν έως και 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην τρίτη μας θητεία, η οποία ε, θα εκπνεύσει τον Οκτώβριο του 2014 παράλληλα και με την λήξη της Επιτροπής Βαρόσο, της δεύτερης Επιτροπής Βαρόσο για πρώτη φορά εξετάζουμε το πόσο ή πώς μπορεί η δημόσια διοίκηση στα κράτη-μέλη να εργαστεί πιο αποτελεσματικά και πώς μπορούν να υλοποιηθούν σε επίπεδο κρατών μελών και δημόσιας διοίκησής τους οι περιορισμοί του γραφειοκρατικού φόρτου, όπως θα λέγαμε και θα με καταλάβουν καλύτερα στους Γερμανοί, ένα είδος μελέτης πίζα για να δούμε ποια είναι η δημόσια διοίκηση που έχει καλύτερα αποτελέσματα. Και έτσι να πούμε ότι να κοιτάξτε εδώ υπάρχει ένα ζήτημα δεν είναι γνωστό ακόμη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι και πώς υλοποιείται και αυτό πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Το έχει πει και ο κύριος Βαρόσο. Με συγκεκριμένη δουλειά λοιπόν όπως αυτή που κάνουμε σε αυτή την τρίτη θητεία και όπως είπα είμαστε ε, μια ομάδα υψηλού επίπεδου, εργαζόμαστε μόνο ε, επιτιμή, δεν έχουμε δηλαδή αποφασιστικές ή καθοριστικές αρμοδιότητες και μπορούμε απλώς να διατυπώσουμε συστάσεις. Αλλά το έχω πει και από την πρώτη φορά και πιστεύω ότι ο κυριότερος στόχος πρέπει να είναι όχι η ανάληψη του ενός ή του άλλου μέτρου, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας στις Βρυξέλλες. Και πρέπει ο νέος κανόνας να είναι ότι δεν είναι υποχρεωτικό να αριθμίζεται οτιδήποτε είναι δυνατό να αριθμιστεί νομοθετικά σε επίπεδο Βρυξελών. Χρειαζόμαστε μία τριπλή διασφάλιση. Θα σας το πω με μια εικόνα. Μπορεί να έχουμε ένα παντελόνι και να θέλουμε να το ασφαλίσουμε με μια ζώνη. Ε, εάν κάθεστε ε, σε μια καρέκλα και σπάσει ξαφνικά η ζώνη σας, πρέπει να φοράτε τυράντες για να το κρατήσετε, να μπορέσετε να σηκωθείτε ψηλά. Και αν τυχόν φοβάστε και να σπάσουν και οι τυράντε, το λάστιχο τη τυράντα, ε, να έχετε και μία παραμάνα να κρατάει με το πουκάμισο το παντελόνι για να μην πέσει. Αυτό λοιπόν θα ήταν μια τριπλή ασφάλεια, όπω διασφάλιση, όπω θα την ήθελα εγώ, για την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό νομίζω ότι θα σήμαινε μια τριπλή επαλήθευση ότι χρειάζεται μια ε, ευρωπαϊκή ρύθμιση μόνο για συγκεκριμένα ζητήματα. Να μην πούμε δηλαδή, να μην λέμε δηλαδή ότι πρέπει η πίτσα Ναπολιτάνα που θα πουλάει η πιτσαρία από το ένα άκρο της ε, Ευρώπης έως το άλλο θα πρέπει να έχει ε, ύψος τόσα εκατοστά ή χιλιοστά διάμετρο τόσα ή τόσα και δεν ξέρω τι άλλη λεπτομέρεια διαφορετικά δεν δικαιούται να φέρει το όνομα πίτσα Ναπολιτάνα ή το, ή το αλυσιδάκι που βάζουμε στην πιπίλα των μωρών. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα κοιτάξουμε με ένα διαφορετικό μάτι. Και γι' αυτό χαίρομαι. Το είδατε νομίζω και στο Στρασβούργο. Είχατε την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης του Προέδρου Μπαρόζο, όπου στην τελευταία σελίδα εγώ είδα το πιο σημαντικό και ενδιαφέρον ζήτημα. Πολύ καλή ομιλία, δεν νομίζω όμως να έμεινε κανείς άναυδος από το μεγαλείο τη, Ωστόσο στο τελευταίο κομμάτι υπήρχε, στο τελευταία σελίδα υπήρχε η ιδέα ότι πρέπει η ευρωπαϊκή ιδέα να αξιοποιείται οπουδήποτε υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να φέρει την ευρωπαϊκή ιδέα. Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι κάθε ευρωπαϊκός κανονισμός, ευρωπαϊκή διάταξη ήταν περσέ αυτόνομα, αυτή καθεαυτή, και μια καλή ρύθμιση. Μέχρι τώρα και αυτό ήταν το πνεύμα της ε, παλαιάς σχολής. Τώρα όμως αυτό αποτελεί παρελθόν. Ο, Επίτροπος, ο πρόεδρος Βαρόσο και στις 2 Οκτωβρίου μάλιστα το 2013 με το πρόγραμμα REFIT παρουσίασε αυτή την αλλαγή τάσεως και στάσεως και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε μια ανάλυση του συνολικού δικαιικού πλησίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζει για κάθε τομέα πολιτικής που μπορούν να απλουστευθούν οι διατάξεις. Αυτό είναι τεράστιο έργο. Δεύτερον, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει σε αποχή, παράληψη ρύθμισης υποβολή νομοθετικών προτάσεων, όπου αυτό δεν χρειάζεται. Και έτσι απορρίπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτοβουλίες νομοθετικές όπου δεν χρειάζονται. Φεριβίν, ε, τι παπούτσια πρέπει να φοράνε οι κομμωτές και οι κομμωτριές μέσα στο χώρο εργασίας τους. Δεν πρέπει να είναι βέβαια θέμα ευρωπαϊκής ρυθμίσεως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει επίσης, όπως ανακοινώνει ο πρόεδρος Μπαρόσο, να εξετάσει τι είδους διατάξεις και σε ποιο βαθμό πράγματι υλοποιούνται οι ευρωπαϊκές διατάξεις στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Και εδώ ακριβώς μας ενδιαφέρει και εμάς ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο το εάν, αλλά και το πώς γίνεται αυτή η υλοποίηση. Και σημειώνω τα λόγια του Προέδρου της Επιτροπής ότι 74% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει πολύ γραφειοκρατία, και ότι πρέπει να ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο με τα μεγάλα ζητήματα και να απέχει από τη ρύθμιση των ίσονος σημασίας ζητημάτων. Σε αυτό συμφωνώ, συμφωνούμε και νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται και στις ανησυχίες και τις ευαισθησίες των Ευρωπαίων πολιτών. και αποτελεί ταυτόχρονα μέτρο της επιτυχίας μιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Από αυτό θα εξαρτηθεί η ευρωπαϊκή πολιτική, από αυτό, είτε είναι ο Σούλτ είτε είναι ο Γιούγκερ, θα κριθεί και ο νέος πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και βεβαίω με όλα τα μεγάλα, με όλες τις μεγάλες ιδέες και τα οράματα που ακούμε από τον Γιούγκερ και τον ε, Σούλτς, ξέρουμε ότι πάνω απ' όλα θα κριθούν από το εάν επιτύχουν να φέρουν αποτελέσματα στο ζήτημα της γραφειοκρατίας. Εγώ, για να ολοκληρώνω, έχω μεγάλα, ε, μεγάλες προσδοκίες ύστερα από τόσα χρόνια ε, δουλειά στην ομάδα υψηλού επίπεδου αλλά και από την πολιτική μου διαδρομία, θεωρώ ότι θα πρέπει και η δημόσια διοίκηση να εμπεδώσει αυτήν την τοποθέτηση και τις ε, εξαγγελίες του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να εγκαταλείψει μία στάση η οποία έχει οδηγήσει στην στο χαρακτηρισμό του, Ευρωπαίου... του Ευρωκράτη, όπως λέμε, με τόσο αρνητικά χρώματα. Έτσι λοιπόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει βεβαίως να παίξουν λίγο μικρότερο ρόλο. Δεν λύνεται δηλαδή το πρόβλημα της γραφειοκρατίας με την υπαοβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Του αντίον θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συμμετέχει και στο διάλογο για το τι σημαίνει ένα νομοθέτημα, τι συνέπειες μπορεί να φέρει και τι είδου γραφειοκρατία. Και μπορώ να σας πω, το Γερμανικό Κοινοβούλιο το θέμα αυτό ε, δεν το μελετά πολύ διεξοδικά το ζήτημα δηλαδή των συνεπειών ενός μιας ρυθμίσεως όπως νομίζω και τα περισσότερα από τα εθνικά κοινοβούλια. Ωστόσο πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μπορέσει, το έχετε επιτύχει εσείς να προχωρήσει σε μια αξιολόγηση τέτοιου, τέτοιων συνεπειών και κόστους και θα πρέπει να ακολουθήσει το επόμενο βήμα και να φροντίσουν τα τρία θεσμικά όργανα να προβαίνουν σε μια ανεξάρτητη και σοβαρή αξιολόγηση των συνεπειών κάθε νομοθετήματος και ελπίζω αυτό, αυτή την αξιολόγηση που χρόνια τώρα την ζητά και την επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να τη δούμε να υλοποιείται. Ε, θα ήθελα επίσης πολύ προσεκτικά να πω ότι όλο και περισσότερο αισθάνομαι ότι με βλέπουν σαν έναν διαμεσολαβητή για κάθε είδους αίτημα και ανησυχία ε, για το θέμα της νομοθεσίας και της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω κι εγώ ασχοληθεί πολύ με τα θέματα αυτά. Έχουμε εξετάσει λοιπόν διάφορες προτάσεις. Έχουμε συλλέξει και προτάσεις offline όπως ονομάζονται και τις έχουμε συμπεριλάβει στις συστάσεις της ομάδας μας για να τις διαβάσουμε στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας έχει απασχολήσει πολύ το θέμα αυτό και θα ήθελα με ένα παράδειγμα να σας πω με ένα, για έναν Γερμανό πολίτη ο οποίος τώρα ζει στην Ισπανία και ο οποίος ε, μας εξήγησε πόσο δύσκολο ήταν ε, γραφειοκρατικά το αυτοκίνητό του που είχε αγοράσει στη Γερμανία να το μεταφέρει και να το καταχωρήσει στην Ισπανία. Μα έχουμε κάθε χρόνο 3,5 εκατομμύρια πολιτών ή και επιχειρήσεων που μεταθέτουν την έδρα τους ή την κατοικία τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Και χρειάζεται να ε, λαμβάνουν ε, τα νέα χαρτιά, τα νέα στοιχεία και τις ε, άδειες ή τα, τα, την τεκμηρίωση για την εγκατάσταση και τη διαμονή κτλ. Μα αυτό θα έπρεπε να ισχύει μια διαπαντός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα να υπάρχει μία λύση με μία υπηρεσία στην οποία θα μπορούμε να απευθυνόμαστε με έναν Ευρωπαίο εκπρόσωπο για την ε, αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, πράγμα για το οποίο εγώ δεν θα ήμουν υποψήφιος, ίσως κάποιος ευρωβουλευτής να μπορούσε να καλύψει θέση αυτή πιο πολύ πιο επιτυχώς και ο οποίος θα μπορούσε και με την δικτύωση που χρειάζεται στις Βρυξέλλες να ε, στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια για τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου. Γιατί χρειάζεται ένας σαφής στόχος και ένα σαφές καθαρό αποτέλεσμα στον αγώνα αυτό για την κατάργηση της ε, γραφειοκρατίας. Γιατί δεν μπορούμε να το επιτύχουμε όπως ακριβώς το επιθυμούν οι πολίτες. Διότι πολύ συχνά αντί να καταργείται η γραφειοκρατία ενισχύεται. Και εδώ χαιρετίζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια ζητεί την κατάργηση της γραφειοκρατίας. Αυτό το ακούμε όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα και πριν από τις ευρωεκλογές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τρία λοιπόν θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο, μπορούν να κάνουν μια δήλωση πριν από τις ευρωεκλογέ για να απευθυνθούν στους πολίτες και να εξηγήσουν αυτή την προσπάθεια. Αυτό θα ήταν νομίζω πολύ σημαντικό. Και αυτό επίσης θέλω να υπογραμμίσω ότι πρέπει να γίνει πιο γρήγορη η Ευρώπη. Να εργάζεται πιο γρήγορα. Ένα παράδειγμα έχουμε από τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το γνωρίζετε πολύ καλά, την ε, κατάργηση της υποχρέωσης για, τις ε, μικρές, για τα μικρά φορτηγά όταν διανύουν απόσταση μέχρι 100 χιλιόμετρα να χρησιμοποιούν ψηφιακό ταχογράφο. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις που δεν είναι αποδεκτές. Πρέπει η Ευρώπη, πρέπει οι Βρυξέλλες να ρυθμίσουν τα μεγάλα ζητήματα, τα δε ίσονο να τα αφήνουν στο εθνικό, το περιφερειακό, το τοπικό επίπεδο. Οι κάτω χώρες τον Ιούνιο του 2013 κατέγραψαν σε μια λίστα επικουρικότητες, όπως τη λένε, τον κατάλογο των προτάσεων που όπου μπορεί να ασκείται η αρμοδιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκείνων όπου Υπάρχουν επιφυλάξεις και διατυπώνονται από τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, στη συνεδρία του Συμβουλίου. γιατί θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραλείψει την ανάληψη νομοθετική πρωτοβουλία για τα θέματα αυτά. Οι Βρετανοί, με την έκθεση Κάμερον όπω ονομάζεται, προχωρούν ακόμη περισσότερο προ την απορρίθμιση σε στυλ Θάτσερ καταργώντας ευρωπαϊκές προδιαγραφές ακόμη και στο εργατικό δίκαιο, την προστασία εγγύων γυναικών ε, από τις απολύσεις και το καθεξής. Αποτέλεσμα, ο Ντέιβιτ Κάμερον που έφερε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο και δεν συζητήθηκε, γιατί ξέρετε βέβαια το υπόβαθρο, ξέρετε τι είδου προτάσει είχαν διατυπωθεί, τροποποίηση των συνθηκών, δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2017. Όλα αυτά λοιπόν έχουν τη σημασία τους για το θέμα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει, δηλαδή το smart regulation όπως το λέμε, την ευφύ νομοθετική παρέμβαση και ρύθμιση. Και είμαι πεπισμένος ότι η νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το smart regulation, ευφύης ρύθμιση, είναι κλειδί για το μέλλον, είναι εκφαντικό άλμα. Και σε έναν κόσμο περίπλοκο όπως ο δικός μας, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην πολύ βασική ιδέα της απορρίθμισης σε στυλ Μάργαρη Θάτσερ. Δεν θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται η ρυθμίση και παραμένει η ανάγκη για ρυθμίση σε κάποια ζητήματα, αλλά όσο το δυνατόν λιγότερο επαχθός. Και γι' αυτό υποστηρίζω αυτή τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί είμαι πεπισμένος ότι θα συνεχίσει το δρόμο αυτόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι θα αποδειχθεί στην προσπάθεια αυτή κατά πιο φιλόδοξο ακόμη τρόπο και ότι θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και τον Απρίλιο και τον Μάιο και ίσως και τον Μάιο με τις ευρωεκλογές να δούμε τα, τις προσδοκίες των πολιτών που είναι πολύ πιο υψηλές από ό,τι πριν από 5, 10, 15 χρόνια ε, ελπίζω λοιπόν ότι τα θέματα αυτά θα απασχολήσουν το δημόσιο διάλογο και στις κατοχώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα κρατημέλη ασφαλώς. Και το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει κάθε πρόβλημα που ε, ε, ανακύπτει στην Ευρώπη να είναι να ρυθμίζεται από την Ευρώπη. Όπως είπα, η πίτσα Ναπολιτάνα δεν πρέπει να ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επικουρικότητα πρέπει να επανεξεταστεί και να επανατεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ο δρόμος για τις Βρυξέλλες δεν μπορεί να είναι μονόδρομος. Με αυτά ελπίζω και για τα επόμενα πέντε χρόνια να σας έχω βοηθήσει και θα έλεγα μάλιστα ότι αν είναι να κάνω ένα πράγμα και μόνο θα, να, θα, θα ήθελα να μπορέσω να συμβάλλω στην αποδοχή της Ευρώπης από τον πολίτη γιατί είναι υπερβολικά αμαυρωμένη η εικόνα της και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Well, thank you very much indeed, for... Ευχαριστώ κύριε Στόιμπερ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Αυτό που κάνετε, όπως είπα στο ξεκίνημα, η ποιότητα του διοικητικού βάρους ε, είναι σημαντική για την Επιτροπή μας. μία από τις ε, παρατηρήσεις αφορούσε τη μετακίνηση από χώρα σε χώρα αυτοκινήτων και την αλλαγή πινακίδες. Σήμερα θα ψηφίσουμε το θέμα αυτό και να σας πω ότι δεν είναι θέμα της Κομισιόν μόνο, γιατί στην περίπτωση αυτή οι προσπάθειες, οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις εμποδίζουν την πραγματικότητα, γιατί φοβούνται μήπως χάσουν ε, φόρους και ζητούν και μελέτη επιπτώσεων και ξανά μελέτη επιπτώσεων. Εγώ έστειλα μια επιστολή πιο έτσι, πώς το πει σκληρή από ό,τι συνήθως κάτι μέλη λέγοντας ότι αν είχαν κάνει πριν από 18 μήνες μελέτη αντικτύπου, πριν την πρόταση, θα... δεν θα χάναμε το χρόνο μας. την άλλη φορά που θα συναντήσει στο Συμβούλιο θα σου δώσω και ένα αντίγραφο για να ξέρει την απογοήτευσή μα. Υπάρχουν πολλέ ερωτήσει από τα μέλη. Έξι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Μαζί θα ακούσουμε τις... Μαζί θα απαντήσετε, ενιαία θα απαντήσετε. Κόσσνικ, Νίξ, Φαμπ, Στάιλερ, Βάιλερ, Ρούλε, Κρόιτσμαν και Κορία Ντεκάμπος. Κάποιο άλλο. Όλοι δηλαδή στην ουσία. έχουμε μια καλή αντιπροσώπευση όλων των πλευρών. Κύριο Κόσνικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συναντηθήκαμε το 9 και το 10 κύριε Στόιμπερ, δεν ξέρω αν θυμάστε. Τσέχος είμαι. Εξ αρχής ε, στην ομιλία σας μας είπατε ότι μπορεί να ρωτάει κάποιος γιατί τρώμε δύο μέρες τη βδομάδα για το θέμα αυτό. Εγώ είμαι επικεφαλής σε ένα think tank στην Τσεχία που ασχολείται με το διοικητικό βάρος και γνωρίζουμε γιατί είναι σημαντικό και γιατί αφιερώνουμε χρόνο γι' αυτό. Υπάρχει και καλή και κακή γραφειοκρατία. Για να λειτουργεί σωστά η Ένωση, τα κράτη και οι περιφερειές χρειαζόμαστε καλή γραφειοκρατία. Ρωτώ λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά ότι το μεγάλο ζήτημα είναι ποιος είναι επικεφαλής της διοίκησης, η ισχύς, η εξουσία που έχει η εποπτεύουσα αρχή. Δεν πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια ο πολιτικός λόγος Επιτροπής άλλαξε κάπως. Ακούσαμε συχνά τον κύριο Μπαρόζο, ο οποίος μιλούσε με ενθουσιασμό για την ανάγκη να χτυπηθεί η γραφειοκρατία, αλλά τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια αυτό οδήγησε σε νέα γραφειοκρατία με καινούριου κανονισμούς. Η ερώτησή μου είναι, δεν θα έπρεπε η Νέα Επιτροπή να προσπαθήσει να χτυπήσει τη γραφειοκρατία όχι μόνο στο ξεκίνημα της θητείας της, αλλά σε όλη την περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Στόιμπερ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας να μας μιλήσετε σήμερα. Τέσσερα χρόνια δουλειά πίσω μας και η έκθεση που μας παρουσιάζεται σήμερα νομίζω δείχνει ότι υπάρχουν επικρίσεις βεβαίως για την ευρωπαϊκή νομοθετική δραστηριότητα αλλά και ότι υπάρχουν και θετικά μηνύματα πώς αλλάζει προς την ορθή κατεύθυνση ό,τι χρειάζεται να αλλάξει. Ε, το 25% για την υποχρέωση ενημέρωσης ε, των επιχειρήσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία, το έχουμε καταγράψει και τα μέσα μαζικής ε, ε, ενημέρωσης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβάλλουμε και εν ώψη των ευρωεκλογών και με αυτά που είπατε νομίζω καθίσταται σαφές ότι εν τέλει η αποδιάρθρωση της γραφειοκρατίας έχει πολιτική σημασία και πολιτική διάσταση και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα ε, όλες οι πολιτικές ομάδες έχουμε ζητήσει και με τη σημερινή έκθεση για τα ευρωπαϊκά τελωνία του κυρίου Κάμπος έχουμε τονίσει ότι πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολικές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, όπως άλλωστε σε όλα τα θέματα. Εγώ αναφερθήκατε μάλιστα και εσείς στον κύριο Μπαρνιέ ε, και την έκθεση Single Market Governance που είχα αναλάβει ε, και που επέτυχε απόλυτη ομοφωνία εδώ για το ζήτημα της υλοποίησης των ευρωπαϊκών ε, προδιαγραφών, ευρωπαϊκών διατάξεων και το ζήτημα ότι η οι δημόσιες προμήθειες στη Γερμανία που ήταν μήλων της έρηδος για χρόνια μεταξύ Ευρώπης και τοπικών αρχών έχει κολλήσει λίγο πολύ στην κακή υλοποίηση από τα κράτη-μέλη της υφιστάμενης νομοθεσίας. Εδώ νομίζω ότι ε, πολύ συχνά κατηγορούμαστε για πράγματα για τα οποία δεν φέρουμε την ευθύνη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και εσείς, αν μου επιτρέπετε να υποβάλω την ε, σύσταση, να συζητήσετε ε, στη Γερμανία και αλλού σε τοπικό επίπεδο δηλαδή. Επίσης, για, τα... για τις μικρορυθμίσεις όπως το αλυσιδάκι της ε, πιπίλας ε, και τα ταχόμετρα που αναφέρατε ή η πίτσα. Να σας πω εγώ ζω σε μια περιοχή που είναι γειτονική με την Ελβετία, είναι όμορη με την Ελβετία. Ε, λοιπόν από την Γερμανία ο πιτσαδόρος δεν μπορεί να πάει να παραδώσει πίτσα στην άλλη μεριά των συνόρων διότι δεν ανταποκρίνεται στις ελβετικές προδιαγραφές ε, η πίτσα αυτή. Ελπίζω τουλάχιστον μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας να είμαστε σε θέση να το επιτύχουμε αυτό, να μην έχουμε δηλαδή τις προδιαγραφές ως εμπόδιο μπροστά μας, όπως συμβαίνει με την Ελβετία. Το ίδιο και για τα ιδιωτική τους αυτοκίνητα και την καταχώρησή τους ε, ε, στα Μητρώα σε μια άλλη χώρα. Αυτό σημαίνει smart regulation βεβαίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ακόμα πιο σοφό θα ήταν το smart deregulation, η απορρίθμιση, η ευφύης, η οποία θα μείωνε τι ε, ρυθμίσεις που επιβαρύνουν του πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και για την ε, απορρίθμιση επίσης. Τώρα η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Δόκτωρα Στόιμπερ, για μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Χαίρομαι που θίξατε το σημείο σχετικά με τον ορισμό του διοικητικού φόρτου, διότι ως αντιπρόσωπος του κόμματος των εργατικών, όταν μιλάμε για αυτό το θέμα, ε, έχει να κάνει με την αφαίρεση των δικαιωματών μητρότητας, για παράδειγμα, με το οποίο διαφωνώ. Ε, χρειάζεται ένας ορισμός, γιατί και τα άλλα θέματα που θίξατε είναι σημαντικά για το 25% μείωση. Το θέμα είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό είναι ε, εξαιρετικό στατιστικό στοιχείο, το οποίο θα μπορούσαμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε στις εκλογές. Θα πρέπει να μεταδώσουμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα ήθελα να δείξω το σημείο για την έγκαιρη προειδοποίηση στα Εθνικά Κοινοβούλια ποια εθνικά κοινοβούλια έχουν τα καλύτερα συστήματα σε λειτουργία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον. Όχι μόνο στη σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και με τα περιφερικά. Εσύ, εγώ είμαι από τη Σκοτία, εσείς από τη Βαβαρία. Ε, εδώ μιλάμε για ε, αυτή την ε, καλύτερη ρύθμιση και θα ήταν ε, καλύτερο να έχουμε αυτή τη ρύθμιση και σε περιφερειακό επίπεδο. Ο κύριος Χάρμπουρ έχει παραθέσει με φράδια τις προκλήσεις μας για τα θέματα εγγραφής οχημάτων. Θα πρέπει να βρούμε τις λύσεις και τους τρόπους. Όχι το σύστημα της πίτσας, αλλά το σύστημα της πίζας. Ε, είναι και αυτό ένα πολύ έγκυρο σημείο. Τώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με 20 χώρες για να έχουμε ένα νομοθέτημα αντί 20 διαφορετικά νομοθετήματα και βλέπουμε ότι δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε εδώ τον ε, διοικητικό φόρτο, αλλά να έχουμε καλύτερο διάλογο. Και τέλος, ποιο είναι το μέλλον του οργανισμού σας, πώς θα λειτουργήσει και προς τα που οδεύει. Γιατί αυτό που έχετε κάνει μέχρι στιγμής είναι εξαιρετική δουλειά. Αλλά πώς ποια συνέχεια θα δοθεί, διότι είναι τόσο ζωτική σημασία στο έργο σας. Ευχαριστώ, Κάθριν. Κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα και από μένα, κύριε Στόιμπερ. Η σύντομη τοποθέτηση σας άγγιξε ένα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη πάντως. Λέτε ότι δεν θα αναφέρεστε στα μικρά παραδείγματα. Ναι, αλλά τα μικρά παραδείγματα είναι αυτά τα οποία αμαυρώνουν την εικόνα της Ευρώπης πολλές φορές δίκαια αλλά και πολλές φορές άδικα. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε πιο σαφείς γιατί υπάρχουν ε, κάποια με, ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία επιδιώκουν και γνωρίζουν καλά την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία και δίνουν μια καθαρή και αντικειμενική εικόνα, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα, ακόμα και από τα πολύ σοβαρά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ε, ε, μεταφέρουν εσφαλμένες πληροφορίες. Και στη δική μου την περιοχή, στο ΕΣΕΝ, φαίνεται ε, ότι μία απόφαση η οποία ανήκε στην τοπική κυβέρνηση που είχε να κάνει με την ε, ιδιωτική κατανάλωση του ύδατος, ε, ε, την ίδρυψη δηλαδή, χρεώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τρόπο άδικο. Εμείς λοιπόν εδώ στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς δεν είμαστε η κατάλληλη επιτροπή για να ακούσουμε τις εκκλήσεις σας, γιατί ήδη εδώ και χρόνια επεξεργαζόμαστε μια αντικειμενική, ουδέτερη και λειτουργική προσέγγιση Προσπαθούμε, επί παραδείγματι όπως ξέρετε, και ύστερα από 20 χρόνια συζητήσεις, να βρούμε ε, μία λύση για ένα ενιαίο φορτιστή για τα κινητά τηλέφωνα. Προσπαθούμε. Επίσης, ακούω ότι και η γερμανική ε, υπηρεσία ελέγχου των διατάξεων έχει αποδηθεί σε μια προσπάθεια για περιορισμό της γραφειοκρατίας, που όμως 10 ε, χρόνια μετά έχει διωγγωθεί αντί να Άρα ο έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Επίσης αναφέρεστε σε μια λογική τοποθέτηση σε μια αντικειμενική και ορθολογική προσέγγιση. Ναι, αλλά πολλά είναι ζητήματα πολιτικών επιλογών και γνωρίζω, όχι στη δική μας την Επιτροπή, αλλά ότι η συνάδελφοι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε προωθήσει ιδιαίτερα την ιδέα του οικολογικού σχεδιασμού, την είχε εγκρίνει εκτός από κάποιους συντηρητικού. Εμείς δεν είχαμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό γιατί είχαμε άλλα ζητήματα, αλλά και από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ξέρω ότι έχουμε μια σειρά από διατάξεις ε, σχετικές με την κοινωνική προστασία, προστασία παραδείγματι από την χορύπανση στο χώρο εργασίας που ε, είχα εγώ ιδιαίτερα παρακολουθήσει με τη Helen John Smith και που ε, όμως ε, από τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης στη Γερμανία παρουσιάστηκαν με τελείως ασφαλμένο τρόπο και πέρασαν δύο χρόνια για να περάσει, ενώ η αρχική απόφαση που είχε ληφθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε λάβει πολύ αρνητική διαφήμιση ή ε, παρουσίαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν δύο χρόνια μετά μπήκε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της Γερμανικής Βουλής, τότε έλαβε εγκομιαστικά σχόλια από τον ίδιο αυτόν τύπο. Ανάλογα με το ποιο ήταν το όργανο το οποίο επεξεργαζόταν δηλαδή το ίδιο νομοθέτημα. Άρα ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωση μεταφέρουν, μεταδίδουν τις ειδήσει. Ναι βεβαίως εν ώψη των ευρωεκλογών είναι απαραίτητο να μιλήσουμε για αποδιάρθρωση και περιστολή της γραφειοκρατίας αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Ευχαριστώ κύριο Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πολύ. Δύο-τρεις τοποθετήσεις από την εμπειρία που έχω συλλέξει αυτά τα χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε πολλούς επιτρόπους, διότι οι επιτροποί, ε, ξέρετε, πρέπει να αποδείξουν ότι κάνουν και τη δουλειά τους, ότι έχουν λόγο ύπαρξης δηλαδή. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αυτά τα οποία έχει να κάνει, αλλά δεν αξιολογεί στη συνέχεια ή δεν ζητείται η αξιολόγηση ε, των συνεπειών του νομοθετήματος όταν έρχεται και περνάει αυτό από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι σε πολλά πράγματα και με τις χιλιάδες τροπολογιών που περνούν ε, από το Κοινοβούλιο επιδεινώνεται ένα νομοθέτημα όταν ρυθμίζονται όλο και πιο μικρές λεπτομέρειες ε, και γίνεται πιο περίπλοκο το νομοθέτημα. Επίσης, στον τριμερή διάλογο που έχουμε ασχοληθεί οι συνάδελφοι και εγώ Έχουμε ξαφνιαστεί από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου που μας είπε ότι δεν υπάρχει παρκής χρόνος για την προετοιμασία των δημοσίων, των διαγωνισμών για τις δημόσιες προμήθειες και ότι κράτη όπως η Γερμανία έχουν ε, πατήσει το φρένο στις διαπραγματεύσεις επίπεδο Συμβουλίου ενώ άλλα κράτη όπως η Πορτογαλία είχαν μπορέσει να προχωρήσουν πάρα πολύ ταχαίως στην ηλεκτρονική οργάνωση όλης αυτής της διαδικασίας και μπορούν να την ολοκληρώσουν συντομότατα. Άρα λοιπόν και πέραν των όσων εμείς εδώ αποφασίζουμε πάνω σε μια οδηγία, έναν κανονισμό, ε, μια οδηγία καλύτερα, πρέπει να ε, περνούν στη φάση υλοποίηση, μέσα στο ε, κράτος μέλος και εκεί θα πρέπει να εξετάσετε πόσοι γραφειοκρατία συνεπάγεται η, το νομοθέτημα της ε, μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Για το κόσμο, επίσης, ο Πομικής Υγητής. Μια μεγάλη ιστορία, πολλή χρόνο θα χρειαστεί, α, πολλές υψηλό το κόστος, να το περιορίσουμε στα 100 ευρώ, γιατί υπάρχουν κράτη που έχουν φτάσει στα, κράτη, κρατήδια καλύτερα που έχουν φτάσει στα 2.000 ευρώ, όλα αυτά από τις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου, διότι πρέπει να τονίσω ότι πολύ συχνά δεν ευθύνεται η Επιτροπή αλλά το Συμβούλιο για όλα τα προβλήματα. Η κυρία Ρούιλε. Κύριε Στόιμπερ, ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Σε πολλά ζητήματα έχετε δίκιο η επικουρικότητα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μελετήσει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το, Ευρωπαϊκό, το νέο κοινοβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές. Ωστόσο πρέπει να πω ότι σε κάποια ζητήματα θα διαφοροποιηθώ γιατί είχα παραδείγματι από το Δημοτικό Συμβούλιο, τοπικό συμβούλιο της ιδιαίτερης μου πατρίδας ότι τον απόϊχο ότι είναι υπερβολικά πολλές ε, οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ελέγχους και υπερβολικά πολλοί έλεγχοι. Από την άλλη ακούμε για την Ελλάδα Φερρυπίν ότι δεν είναι αρκετοί έλεγχοι και ότι σε αυτό οφείλονται κάποια προβλήματα. Ε, λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ούτε μπορούμε όλα να τα λύνουμε με μία, με μία μονοκοντιλιά. Ε, η επικουρικότητα ίσως είναι η λύση, αλλά πρέπει να δούμε και ότι πίσω από την κάθε ρύθμιση κρύβονται κάποια συμφέροντα και εσείς ως Πρωθυπουργός της Βαβαρίας θα θυμάστε ίσως ότι υπήρχε ε, μία ρύθμιση στη Γερμανία, έχει απαιτήσει καλύτερα η Γερμανία μία ειδική ρύθμιση που αφορούσε τις ανεμόσκαλες που χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες. Ε, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Ε, είναι κάτι που χρειάζεται πράγματι η Ευρώπη και ταυτόχρονα είμαστε θέση να λέμε με ειλικρίνεια ότι υπάρχουν και συμφέροντα. Και στην απορρίθμιση ακόμη. Η ιδέα για την απορρίθμιση στο Κοινοβούλιο δείχνει, ε, δείχνει ότι πίσω υπάρχουν κάποια κριτήρια. Πίσω από κάθε απελευθέρωση που σημαίνει και απορρίθμιση ταυτόχρονα το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα το επιδιωκόμενο. Φερρυπίν τηλεπικοινωνίες. Άρα, ναι, είναι ζήτημα η κατάρριξη της γραφειοκρατίας, ο περιορισμός του γραφειοκρατικού φόρτου, αλλά δεν μπορούμε να εξαντλούμε όλο τον προβληματισμό μας σε αυτόν. Ευχαριστώ κύριο Κορέα Ντεκάμπος, μετά Λόκεγκαρτ. ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Στόιμπερ, Ευχαριστώ που μας εκφράσατε τη θέση σας. Μια πολύ πλούσια παρουσίαση που μας επιτρέπει να δούμε και τα δικά μας προβλήματα. Τρία βασικά ερωτήματα. Δεν είναι ότι θέλω να αφώσω τη γραφειοκρατία, αλλά η γραφειοκρατία είναι η βάση του φορολογικού συστήματος. Κανένα κράτος δεν μπορεί να αγνοήσει τη γραφειοκρατία. Δεν δημιουργείται στις Βρυξέλλες. Τα κράτη-μέλη θέλουν γραφειοκρατία γιατί είναι η δομή που εισπράττει. Επίσης, για μια... Ε, χρειάζεται γραφειοκρατία για μια κουλτούρα συμβιβασμού που είναι αναγκαία στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και ε, δεν έχουμε απόλυτη πλειοψηφία ενός κόμματος, άρα πηγαίνουμε σε συμβιβασμούς και άρα η νομοθεσία είναι πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη και ενδεχόμενα πιο απαιτητική γραφειοκρατικά. Εγώ δεν είμαι απεσιόδοξο. Αυτό που έγινε τα τελευταία πέντε χρόνια στην, υλοποίηση, στην ολοκλήρωση τη ενία αγορά είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να θυμίσω απλά ότι το ότι υπάρχει σήμερα τακτική δημοσίευση όλων των ενσωματώσεων ε, ενός νομικού κειμένου από τα κράτη-μέλη, όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και με ποιοτικά αποτελέσματα. Πώς γίνεται αυτό αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Κατόπιν, για την έξυπνη νομοθεσία, το smart regulation. Θέλουμε όλα τα νομοθετικά κείμενα να όχι μόνο αφορούν το, την προστασία του περιβάλλοντος ή την ισότητα αλλά όλα να περνούν το τεστ του Smart Regulation. Εμείς δημιουργήσαμε μια γενική διεύθυνση τώρα μόνο για, τον αντίκτυπο, για την αξιολόγηση του αντικτύπου ενός νομοθετικού κειμένου. Δεν αρκεί η μελέτη αντικτύπου που έχει το νομικό κείμενο και παρουσιάζει η Επιτροπή. Η Επιτροπή θέλουμε μια ειδική γενική διεύθυνση εδώ για αυτό το θέμα. Και μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και συγκρούσει. Ωστόσο, η γραφειοκρατία δημιουργείται πάντα εκεί που αναμενόταν λιγότερο να δημιουργηθεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Στόιμπερ για την παρουσίασή του. Θα είμαι σύντομος γιατί ήρθα καθυστερημένα. Και έχασα ένα κομμάτι από την ομιλία σας. Εμείς οι πολιτικοί ε, λέμε συνέχεια για λίγοι ε, ε, γραφειοκρατία και περισσότερη δημοκρατία. Δεν είναι παράδοξο ότι όσο περισσότερη δημοκρατία αποκτάς τόσο μακρύτερες διαδικασίες έχεις. Υπάρχει ένα παράδοξο λοιπόν με την σχέση δημοκρατίας-γραφειοκρατίας. Εσείς πώς τα λέτε, πώς τα βλέπετε, θεωρείτε ότι υπάρχει αντινομία, θέλετε ένα ανοιχτό κοινοβούλιο με ανοιχτές διαδικασίες και περισσότερη γραφειοκρατία. Πολύ ενδιαφέρουσες και δύσκολες ερωτήσεις. Θα δώσω στον κύριο Στοίμπερ το λόγο για να απαντήσει σε όσες περισσότερες μπορεί, το συντομότερο δυνατό βέβαια, αλλά δεν μπορώ να τον αγνοήσω. Ευχαριστώ πολύ. Και ξέρω ότι έχετε πολύ περιορισμένο χρόνο στη θέση σας. Είναι όμως ε, θεμελιώδη τα ερωτήματα. Δώστε μου λοιπόν μερικά λεπτά ώστε να δώσω στο βαθμό που μπορώ τις απαντήσεις. Πρώτο σημείο. Θέλω να καταστήσω απόλυτα σαφές ότι το δικό μου αίτημα είναι και το δικό σας αίτημα εν γέννη και να πω ότι η Ευρώπη είναι ένα συναρπαστικό εγχείρημα, μια συναρπαστική ιδέα, ένα μοναδικό στον κόσμο εγχείρημα και τώρα που αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη κρίση με την Ουκρανία και πάλι επανέρχεται βέβαια στην ε, επικαιρότητα, στο φως των προβολέων, ότι θέλουμε να είναι σε θέση η Ευρώπη να διατυπώνει μία ιδέα και μία γνώμη σε σχέση και την με τη Ρωσία. Χαίρομαι που ένας Γάλλος, ένας Γερμανός, ένας Πολωνός, ένας Ούγγρος υπουργός, κάθονται να συστήσουν για να προσπαθήσουν να διατυπώσουν μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση και θέση εναντί της Ρωσίας. Αυτό σημαίνει ακριβώς και απτά η Ευρώπη. Από την άλλη, και πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, και εγώ προσωπικώς και δεν έχω καμία άλλη φιλοδοξία, η δική μου πολιτική αεροδρομία έχει κλείσει, την έχω πίσω μου και την Ευρώπη μπορώ από ιδεολογική ε, προσέγγιση να τη δω, όχι για λόγους πολιτικού σχεδιασμού και υπολογισμού. Και να πω ότι με εξοργίζει το ότι μπορεί κανείς να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να αντιμεταστρέψει προς το ένα ή το άλλο θέμα δίνοντας με ένα, με ένα μεγάλο τίτλο το, την ιδέα ότι η τάδε ρύθμιση επιβαρύνει πολύ τους πολίτες και ότι είναι περιττή και ότι ενοχλεί και όλα αυτά. Η Ευρώπη, και αυτή είναι η πολιτική μου εμπειρία, ισοδυναμεί με τα θεμέλια του ευρωπαϊκού ιδεόδους. το να μιλούμε για γραφειοκράτες, ευρωκράτες και όλα αυτά, ωραίες ιδέες, αλλά δεν είναι η γραφειοκρατία μόνο αυτή της Ευρώπης, είναι και αυτή της Ισπανίας ή της Γαλλίας. Δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι στην, ε, στο Βερολίνο φέρει πίνη δημόσια διοίκηση είναι όλο ε, γραφειοκράτες και μια κυβέρνηση υπάρχει όπως η Μέρκελ, όπως ο Κάμερον, όπως ο Ολάντ. Στην Ευρώπη όμως χρεώνονται τα πάντα οι ευρωκράτες που είναι και οι κακοί. Γι' αυτό λοιπόν, και το λέω και πολιτικά, αλλά και με μια σειρά από επιχειρήματα, χαίρομαι που σε αυτή τα, την επταετία, σε αυτά τα 7 χρόνια, μπόρεσα 16 φορές να έρθω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλές φορές στο, κοινοβου, στο Συμβούλιο, επίσης βέβαια και προφανώς σε συνεργασία με την Επιτροπή και επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχω έρθει και έχω συνομιλήσει με τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, τα μεγάλες πολιτικές ομάδες, σοσιαλιστές, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Φιλελευθέρου. Σε όλες, αυτές, σε όλες αυτές τις ομάδες βλέπω ξεκάθαρα τον στόχο και τη βούληση του περιορισμού του γραφειοκρατικού φόρτου. Μπορεί στο ένα ή το άλλο ε, ζήτημα ρύθμιση να υπάρχουν μικροδιαφοροποιήσεις, αλλά ο στόχος είναι κοινό. Και επίσης, όπως λέω, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρέπει να ξανακοιτάξουμε τα θεμέλια και να δούμε φερρυπίν την συμφωνία για το παγκόσμιο εμπόριο. Μπαλή Νοέμβριος, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό στόχο που και πάλι έχει εγγραφεί, που είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και που υπολογίζεται ότι θα εξοικονομήσει ένα δισεκατομμύριο σε δολάρια ε, από την απλούστευση των διατάξεων από τα αφρικανικά κράτη, από εδώ και από εκεί. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει και σε αυτό να συμβάλλει σε ένα μικρό μέρος έστω, σε έναν τόσο περίπλοκο κόσμο, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Αυτό που θέλω να απαντήσω δε στον κύριο Κρότσμαν το είπε ο κύριος Λόκεγκαρτ. Βεβαίως η δημοκρατία βαίνει παράλληλα σε ένα βαθμό με την γραφειοκρατία. Δεν μπορώ δηλαδή να έχω ένα σύστημα δημοκρατικό εάν δεν μπορώ να εξασφαλίσω την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών και άρα να έχει ο πολίτης τη δυνατότητα να ε, την χάνει της ίδιας αντιμετώπισης από το κράτος και άρα να έχει την δυνατότητα και την απέτηση και να υφίστανται όντω οι κανόνε που θα εξασφαλίσουν αυτή την ισότιμη μεταχείριση. Διότι εάν δεν υπάρχουν κανόνε, δημοκρατία δεν μπορεί να υφίσταται. Θα είναι μόνο αυθαιρεσία. Η γραφειοκρατία όμω δεν μπορεί επειδή υπάρχει να μαυρώνει τη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να πετάμε στα σκουπίδια τη δημοκρατία λόγω της γραφειοκρατίας και να λέμε δεν χρειάζεται. Ξέρω ότι και εγώ πολλές φορές έχω αδικαιολόγητα επικρίνει την Ευρώπη. Το ομολογώ. Αλλά εδώ δεν είναι η ουσία του ζητήματος. Η ουσία είναι ότι η Ευρώπη έχει πολλά ακόμα να πει και δυστυχώς οι πολίτες δεν το γνωρίζουν. Πάνω από χίλιους κανονισμούς εκδίδει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. 1.900 οδηγίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά ο πολίτης δεν ξέρει τι εφαρμόζεται σε ποια περίπτωση. Δεν γνωρίζει καλά, δεν ξέρει ποια είναι τα διάφορα επίπεδα της διοίκησης. Θεωρεί ότι τα αποφασίζει όλα η Επιτροπή, ότι αποφασίζει τους νόμους, δεν ξέρει ότι η υλοποίηση γίνεται σε παιδοκρατών κρατών μελών. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα κοιτάξουμε και να αναλογιστούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Αυτή ήταν μια επικεφαλίδα θα έλεγα, μια γενική, ένας γενικός τίτλος και δεύτερον Τσεχική Δημοκρατία. Η νέα Επιτροπή πρέπει να είναι πιο πολιτική. Θα πρέπει να είναι πιο πολιτική οφείλει να είναι πιο πολιτική και παρακαλώ δεν εννοώ ειδικού και εμπειρογνώμονε που έχουν ε, γενικοί διευθυντές και γενικές διευθύνσεις. Χρειαζόμαστε και πολιτικούς εκπροσώπους. Τα σχόλια είναι εκτός μικροφώνου δυστυχώς. Κοιτάξτε να σας πω, έχω την εμπειρία. Δεν υπάρχει οργάνωση ή κυβέρνηση στην Ευρώπη η οποία να δέχεται τέτοιες ε, κατηγορίες και να μην αποκρίνεται όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε ξέρουμε ότι εάν δεν εξασφαλίζουμε την αποδεξιμότητα, την αποδοχή, δεν μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα. Ε, αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το ρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από ε, μία υποπαράγραφο που θα γράψει ένας υπάλληλος ή συνεργάτες. Αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη. Υπάρχει μια σαφής προοπτική. Έχουμε δύο υποψηφίους, τον οποίο ο ένας θα γίνει πρόεδρος της Επιτροπής, ή ο Σούλτς, ή... Όχι, γιατί κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω, πολιτική μου παρατήρηση, ότι αν, θέλει ο ένας το θέλει ο ένας ή ο άλλος αρχηγός κυβέρνησης, έστω και της γερμανικής κυβέρνησης, ε, θα αποφασίσει μονομερός. Όχι. Δεν συμβαίνει αυτό πλέον, δεν περνάει. Ο ένας από τους δύο θα γίνει πρόεδρος επιτροπής. Ο άλλος, εάν γίνει ο άλλος ο οποίος δεν έχει εξασφαλίσει την πλειοψηφία, τότε θα προκύψουν τεράστιες συγκρούσεις. Και είμαι βεβαίως ότι και ο ένας και ο άλλος θα τηρήσουν μια στάση πολιτικά υπεύθυνη και θα είναι υποδειγματική ως πρόεδροι το ένας το άλλος. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι θα πρέπει και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο με το θέμα της γραφειοκρατίας και να πάρει το παράδειγμα των Τσέχων, ήθελα να το αναφέρω αυτό ω συγχαρητήρια και ω έβαινο προ του Τσέχου Ευρωβουλευτέ, γιατί η Τσεχία έχει αποδείξει ένα τεράστιο αγώνα για την κατάργηση του γραφειοκρατικού φόρτου, άνευ προηγουμένου, αλλά πρέπει να ομολογήσω και ταυτόχρονα ότι βλέπω με κάποια απογοήτευση ότι με τη δεύτερη μας θητεία και τις 74 περιπτώσεις της ε, ε, σύγκριση των βέλτιστων πρακτικών για θέματα που υλοποιούν τα κράτη-μέλη και που είχαμε καταγράψει στην έκθεσή μας, περίμενα ότι αυτό θα, προ... θα οδηγούσε σε μια συζήτηση στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα κάθονταν οι Γάλλοι βουλευτές Φερρυπή να πούνε γιατί δεν είναι η Γαλλία πρώτη-πρώτη στη σειρά. Ή θα έλεγε τον Bundestag για ένα λεπτό. Για την πολίτευση δηλαδή. Ένα λεπτό. Εμείς οι Γερμανοί πίσω από τους Εστονούς ή δεν μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικές προκηρύξεις ε, και μπορούν να το κάνουν ε, οι Πορτογάλοι που έχουν φτάσει στο 75% των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για δημόσιες προμήθειες κτλ. Ενώ εμείς ακόμα είμαστε 12% και το 13% οι Γερμανοί που θεωρούμε ότι τα κάνουμε από όλους καλύτερα. Ε, λοιπόν αυτό, εγώ θα περίμενα κυρίες και κύριοι, ότι στα εθνικά κοινοβούλια θα ξεσπούσε αντίδραση και θα έλεγε στην κυβέρνηση ελάτε εδώ καθίστε κάτω γιατί είμαστε σε αυτή την τόσο κακή θέση τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, κοστή. Γι' αυτό λοιπόν αυτή είναι η απογοήτευσή μου. Μέχρι τώρα η Επιτροπή δεν ήξερε πώς μπορεί να υλοποιούνται στο κάθε κράτος μέλος αυτές τις διατάξεις. Τώρα όμως πλέον είναι υποχρεωμένη όχι μόνο να επαληθεύσει εάν ε, ε, μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο, αλλά και πώς μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις που έχουν εγκριθεί στο ευρωπαϊκό. Αυτό δεν σημαίνει περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο και το λέμε κάθε ειλικρίνεια. Ξέρω ότι σας πιέζει ο χρόνος. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να ολοκληρώσω τελευταίο. Το Κοινοβούλιο αφήνει το Συμβούλιο να το πιέζει πολύ. Υποχωρεί πολύ. Και ρωτήσα τον κύριο Φαν Ρόμποε για την ε, γραφειοκρατία. Τι κάνει. Είναι ο Μπαρόσο μπροστά στον ε, Ρόμποε φωτεινό παράδειγμα. Ε, κάντε και εσείς κάτι ως κοινοβούλιο. Και είναι γνωστό αυτά. Σε κάθε σύνοδο κορυφή σηκώνεται το Συμβούλιο και Φαν και λέει Α, γραφειοκρατία υπερπάντων και πρέπει να αντιμετωπίσουμε κτλ. Αλλά το Συμβούλιο το οποίο θα πρέπει πιστεύω να αγωνιστεί πολύ περισσότερο και να εξασφαλιστεί ενιαία θα έλεγα στάση μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής με ένα ανεξάρτητο ενιαίο όργανο το οποίο θα προβαίνει στην αξιολόγηση. Α, ναι, έχουμε το impact assessment. Πολύ ωραία, αλλά αφορά μόνο την Επιτροπή, είναι μόνο αρμόδια Επιτροπή. Και αν προβεί σε ε, οποιασδήποτε τροπολογίες τροποποίηση στο Κοινοβούλιο, δεν καλύπτονται από το impact assessment. Ο, ο, όχι, όχι. Ούτε και το Συμβούλιο. Άλλωστε, λαμβάνονται υπόψη. Έτσι νομίζω ότι θα προχωρήσουμε. Και, τελευταία παρατήρηση. Εγώ, για τη Γερμανία, αλλά εσύ και για όλα τα κρατημέλη, φρόντισα να επαληθεύσω πόσες, πόσα διατάγματα αφορούν τον πολίτη τα τελευταία πέντε χρόνια για τη Γερμανία. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τα άλλα κράτη. Πέντε χρόνια. 21.000 νέα, νέα διατάγματα. Εκ των οποίων το 75% από τις Βρυξέλλες. Οι νομοθετήματα θα έλεγα οι Βρυξέλλες έχουν ε, μπει στο πιο μικρό, στην πιο μεγάλη λεπτομέρεια του καθημερινού βίου του πολίτη. Αποφασίζουν τα πάντα. Ξέρετε ότι η Γερμανία έχει ομοσπονδιακή κυβέρνηση και 16 ε, ομόσπονδα κρατήδια, ε, τοπικές κυβερνήσεις και τα 16 τοπικά κοινοβούλια. Και ε, κάποια στιγμή μου είχε προβληθεί το επιχείρημα ότι τελικά δεν είναι και λίγα αυτά που έχει καταφέρει η Γερμανία, αν μπορεί να έχει ένα λειτουργούν κράτος με τα 16, με τα 16 αυτά κρατήδια και την κεντρική κυβέρνηση κτλ. Ναι, μπορεί, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Και γι' αυτό προχωρώ, ζητώντα συγγνώμη αν δεν απάντησα στι επιμέρους ερωτήσεις, ε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη υπόθεση με μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Την τελική μας έκθεση θα την καταθέσουμε στις 16 Οκτωβρίου με τον Παρόζο, τον ε, ασκούντα μάλλον καθήκοντα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα πολύ μεγάλο έργο που θα ξεκινάει και πιστεύω ότι και ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μπορούσε να λάβει από τον Παρόζο ως σύσταση, ως παρακαταθήκη ε, μια ε, έκθεση ολοκλήρωση των εργασιών της προηγούμενης επιτροπής όπου θα έλεγε ότι να εμείς έχουμε κάνει αυτό και αυτό και σας δίνουμε την παρακαταθήκη για να προχωρήσετε με ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση και να διερευνήσετε χάρη στο πρόγραμμα REFIT όλο το νομικό πλαίσιο, να το αναλύσετε και αυτό βέβαια και η Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο, ίσως λιγότερο το Συμβούλιο. Εάν αυτό συνέβαινε λοιπόν σε όλα τα κράτη, γιατί από τα 28 κράτη μόνο 6 έχουν προβεί σε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση συνεπειών. Η Βρετανία, η Ολλανδία, οι κατοχώρες, η Γερμανία, η Σουηδία και η Τσεχία. Πέντε διορθώνω. Τα λοιπά κράτη διατηρούν μια πολύ άνηση εικόνα, χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις ως προς την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και χρειαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε την πολύ αρνητική ε, εικόνα της Ευρώπης, την υπερβολικά αρνητική εστίαση στην Ευρώπη και θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία να γίνει ο δημόσιος διάλογος με όρους αντικειμενικούς και ουδέτερους, με όλους τους ε, σημαντικούς φορείς, ώστε να ρυθμίζονται τα σοβαρά ζητήματα. Όχι τα μικροπράγματα όπως η γλόμπη ε, οικονομίας, οικονομικές λάμπες, λαμπτήρες, αλλά τα σοβαρά και μεγάλα ευρωπαϊκά θέματα θα πρέπει μόνο να ρυθμίζονται από την Ευρώπη. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ίσως τελευταία φορά που σας καλέσαμε σε αυτή την Επιτροπή. Στις 16 Οκτωβρίου, στην τελική σας ε, έκθεση, αν θα είναι μια τόσο ε, ε, ζωντανή παρουσίαση, ελπίζω να κληθούμε να την παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή και πραγματικά σας χαίρω που χειρίζεστε το θέμα με τόσο δυναμισμό και τόσο ενθουσιασμό και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό το ενδιαφέρον και στο μέλλον για πολλά άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρευρεθήκατε εδώ. Κυρίε um, Κυρίες και κύριοι, όπω βλέπετε, είχαμε μια ζωντανή σύνοδο νωρίτερα. Ε, Αυτοί που ήρθατε αργότερα για την ψηφοφορία χάσατε την αρχή. Ε, η Ρόζα είναι πολύ φωτογενής. Βλέπουμε ότι την ε, οπτικογραφούν αυτή τη στιγμή. κάποιες σύντομες ψηφοφορίες ε, θα έχουμε σήμερα το απόγευμα. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι από την ψηφοφορία της περασμένης εβδομάδας στην Ολομέλεια θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όλα τα νομοθετικά μέτρα θα γίνουν με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυτό κάναμε εξάλλου σε αυτή την Επιτροπή. Αλλά θα γίνουν ονομαστικές ψηφοφορίες. Θα καταγράφονται τα ονόματά σας στην τελική ψηφοφορία, μόνο στην τελική ψηφοφορία και η ονομαστική ψηφορία θα δημοσιευτεί στα πρακτικά της συνεδρίασης. Το λέω για να σας πληροφορήσω. μια ερώτηση. Είναι μια αλλαγή στη διαδικασία ή το κάνουμε πάντα έτσι. Όχι. Ε, δεν κάναμε ονομαστικές ψηφορίες, πάντα κάναμε ηλεκτρονικές στο τέλος κάθε διαδικασίας και καταγράφαμε τις πλειοψηφίες. Αυτή τη φορά όμως θα γίνουν Ορμαστικές ψηφοφορίες θα υπάρχει στο τέλος των πρακτικών ένας κατάλογος με τα ονόματα ε, αυτών που ψήφισαν υπέρ, κατά ή που τήρησαν αποχή. Εάν βέβαια αποφασίζετε να μην ψηφίζετε εναπόκειται σε εσά. Αυτά λοιπόν. Περνάμε στα σημεία της ε, ημερήσιας διάταξης. Πρώτα, ο κύριος Ζουβά, ο εισηγητής δεν είναι εδώ, μου φαίνεται. Ήθελα να προτείνω εκ μέρους του και έχουμε κυκλοφορήσει στα μέλη και οι συντονιστές θα το γνωρίζουν, ότι ε, σας καλούμε να εγκρίνετε ένα διορθωτικό στην οδηγία σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παροχώρησης. Δεν θα επισέλθω στις λεπτομέρειες, τα έχετε μπροστά σας. Έχουμε και την τεχνική ομάδα που τα επεξεργάστηκε με τον ισχυτή και του Σκιώδης και συμφωνούμε ότι αυτό το διορθωτικό πρέπει να γίνει. Είναι μια τεχνική διόρθωση που διασφαλίζει ότι όλα τα παρατήματα και όλα τα άλλα στοιχεία ε, έχουν συμπεριληφθεί σωστά. Θα ήθελα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά επ' αυτού και ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία στο διορθωτικό. Πέραση της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 1 κατά. Το επόμενο σημείο Θέλετε να επαναλάβουμε τη διαδικασία. Πείτε μας πώς έχετε ψηφίσει. not working, then. Mm-hmm. Δεν λειτουργεί. Αλλάξτε θέση, ίσως. Θα καταγράψουμε τη ψήφο σας ε, διαχειρός. ούτε εσείς ψηφίσατε, ούτε το δικό σας μηχάνημα δεν λειτουργούσε. Είναι κανείς άλλος που δεν κατάφερε να ψηφίσει. Α, τα μηχανήματα εδώ δεν έχουν λειτουργήσει εδώ και αρκετό καιρό. Έχουν γεμίσει σκόνη. Θα κάνουμε μια ακόμα δοκιμή. Right. We need to move on Πρέπει να προχωρήσουμε όμως. Ψηφοφορία για την έκθεση του καθηγητού Κορέα Ντεκάμπο, αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό διασφάλιση ορθή εφαρμογή των τελωνιακών και γεωργικών ρυθμίσεων. Θα συζητήσαμε τι τροπολογίε. Αν δεν υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία έχουν εγερθεί από τότε, ε, περνάμε κατευθείαν σε ψηφοφορία. Αν συμφωνεί και ο καθηγητή, α ξεκινήσουμε την ψηφοφορία λοιπόν. Άρχεται. Ε, το, τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 43 ε, τοπολογία υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τοπολογία 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τοπολογία 44 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τοπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τοπολογία 46 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται σαφώς. Και πάμε τώρα στην τροπολογία 9 του εισηγητή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 50, κύριο Σμιτ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 από τον εισηγητή υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 51 με προφορική τροπολογία του Όλε Σμιτ με κείμενο έχει εγκριθεί. Ε, η 51 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 11 καταπίπτει, 12 από τον εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 13 του εισηγητή υπέρ κατά Έγκρινεται επίσης. Τροπολογία 52. Ψηφίζουμε διότι η 51 εγκρίθηκε. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 57 του κυρίου Φόξ. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 72 διότι οι ό, όλες οι άλλες έχουν αποσυρθεί. 72 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τοπολογία 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 74 του κυρίου Ρος υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 78 του κυρίου Ρος υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τοπολογία 77 του κυρίου Σμιτ ως επιπρόσθετη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα είμαστε στη συμβαστική τοπολογία 6 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. τοπολογία 54. Με συγχωρείτε, 84 ε, διορθώνει ο πρόεδρος του κυρίου Σμιτ με προφορική τοπολογία υπέρ. Κατά εγκρίνεται σαφώς. Τοπολογία 17 καταπίπτει. 18 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τοπολογία 19 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά εγκρίνεται. 86 It is linked to these two amendments. All right. So, if this him. if this amendment goes through, normally the other two fall, and this was not correctly All right. Okay. Sorry, there was just having. I was just having. a... Ε, μου έχουν δυστεί κάποιες επεξηγήσεις για την 86 που σχετίζεται με μεταγενέστερες τροπολογίες. Θα εξηγήσω τις λεπτομέρειες εάν υπερψηφίσετε. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 86 του κ. Σμίτ. Κατά. Απορρίπτεται. Άρα δεν χρειάζεται να σας δώσω καμία εξήγηση. Ε, κερδίζουμε και χρόνο. Τροπολογίες 21 και 87 μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Η 8 μαζί με την τροπολογία 96 μαζί. Η συμβαστική 8 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Ε, περιλαμβάνεται και η προφορική τοπολογία Συμβαστική τοπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 από τον εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία 100 καταπίπτει. Τροπολογία 28 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 103, 104 και 105 σε μπλοκ υπέρ κατά εγκρίνονται. 106 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 32 ως επιπρόσθετη υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 33 καταπίπτει. Τροπολογία 3 υπέρ κατά Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36 ως επιπρόσθετη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 ως επιπρόσθετο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα θα κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία για την τελική έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ και μια κατά. Και θα συμπεριληφθεί ο κατάλογος στο τέλος των πρακτικών. Τώρα, πάμε, θα περάσει μάλλον στην επόμενη θητεία της ε, Επιτροπής ΙΜΚΟ και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει καλή πρόοδος αυτής. Έχουμε άλλη μια ψηφοφορία. Um, Έχουμε και μια τελική ψηφοφορία για την απλούσευση της μεταφοράς ε, των ε, μηχανοκινήτων οχημάτων. Και θα καλέσω τον εισηγητή να μας εξηγήσει το πλαίσιο αυτής της ψηφοφορίας. Αλλά θα πρέπει να ε, υπάρχει μια ενιαία ψηφοφορία όλων των 106 τροπολογιών και να ληφθεί υπόψη το έργο που έγινε στις άτπες ε, ομάδες εργασίας κατά τη διάρκεια της ελληνική προεδρίας τον Ιανουάριο, διότι το Συμβούλιο δεν ε, διαπραγματεύεται περαιτέρω. Αποφασίσαμε τουλάχιστον να ε, περιλάβουμε τις υφιστάμενες τροπολογίες στην πρόταση, αν δεν μπορεί να έτσι ώστε να μην παραχωρήσει το Συμβούλιο στην επόμενη θητεία. Κύριε Μάντετς, ευχαριστώ. Θέλουμε μία ενιαία ψηφοφορία ε, εκεί που μείναμε με τον μέρη διάλογο, όλοι οι σκιώδεις ε, συμπεριλαμβανομένου και του εισηγητή ήταν πολύ απογοητευμένοι με την επιστολή του Συμβουλίου που δεν ήθελαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις διότι πρώτα θέλουν να έχουν αντι... Ε, εκτίμηση αντικτύπου. Και αυτό οθήθηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών και όχι τους Υπουργούς Μεταφορών. Το είπε και ο κύριος Στόιμπερ. Είναι ε, ένα από τα θέματα που προκαλούν πολύ μεγάλη απογοήτευση στην Ευρώπη και αν το Συμβούλιο δεν θέλει να πραγματευτεί περαιτέρω είναι κρίμα πραγματικά. Ελπίζω να στηρίξουμε την ενιαία ψηφοφορία, θα έχουμε μια συμφωνία επί πρώτης ανάγνωσης και ελπίζω κύριε Πρόεδρε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια στεναρή δήλωση στην Ολομέλεια τον Απρίλιο όταν θα ψηφίσουμε και ίσως να μελετήσουμε και το ενδεχόμενο να δείξουμε ότι το Συμβούλιο δεν βοηθάει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη στάση του. Σε πρώτη ανάγνωση, δεν υπάρχει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, είμαστε στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης ακόμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης, οι ε, και την Επιτροπή Δουλέψαμε πολύ σκληρά μαζί και νόμιζα ότι είχαμε πλησιάσει πάρα πολύ σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία επί πρώτης ανάγνωσης, διότι είχαμε ε, πετύχει σχεδόν σε όλα όσα είχαμε σφίσει και τελικά απογοητευτήκαμε. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια πολύ δυνατή δήλωση στην Ολομέλεια για να δείξουμε ότι το Κοινοβούλιο ήθελε να έχει καλύτερη λειτουργία στην Ευρώπη και το Συμβούλιο παρεμποδίζει αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ κανείς από τους συντονιστές θέλει το λόγο. Α, η κυρία Γκέπχαρτ. Κάτι που δεν κατάλαβα. Γιατί είναι η διαδικασία. Και δεν ήμουν ενημέρη εκ των προτέρων ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Θα ήθελα να μου πείτε τι είδου συνέπειε φέρνει αυτό που προτιθέμεθα να κάνουμε εδώ. Έχουμε μια σειρά από πολύ καλές τροπολογίες εδώ στην Επιτροπή. Ο κύριος Μάντερς έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τώρα γίνεται μια νέα ψηφοφορία στην Επιτροπή για μια σειρά από τροπολογίες που εν μέρει είναι συμβαστικές με το Συμβούλιο, Συμβασμένο με το Συμβούλιο. Ερωτώ λοιπόν τι σημαίνει αυτό για τη λυπή διαδικασία στη διάρκεια της υπόλοιπης θητείας, όταν θα έχουμε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο ή όταν θα κληθεί το Συμβούλιο να λάβει μια απόφαση. Θα αποτελεί αυτό βάση για νέα εκκίνηση διαπραγματεύσεων. Το Συμβούλιο δηλαδή έχει υποσχεθεί ότι αυτά, εφόσον τα ψηφίσουμε, ισχύουν και δεν τα ξανανοίγει τα θέματα ή τελικά μπορεί και να ανατρέψει ζητήματα τα οποία είναι βασικά για το Κοινοβούλιο. Αυτό θέλω να καταλάβω τι κάνουμε τώρα και τι συνέπειες θα έχει για την περαιτέρω μοίρα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Θες να απαντήσεις εσύ, ναι. Εύλην, είχαμε την επιλογή είτε να περάσουμε στην Ολομέλεια το αποτέλεσμα που ψηφίζουμε στην ΙΜΚΟ σε πρώτη ανάγνωση. Εμείς σαν με τους Σκιώδης ξεκινήσαμε να συζητούμε αυτά που μπορούσαμε να δεχθούμε στην άτυπη, στους άτυπες διαπραγματεύσεις και είπαμε ότι Τη στιγμή που τελειώνουμε τις διαπραγματεύσεις θα ήταν καλύτερο ίσως να δείξουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να συμβιβαστούμε με το Συμβούλιο. Συμβιβασμούς προτείνουμε τώρα. Οι σκιώδεις ηγητές είπαν το συζητήσαμε και συμφωνήσαμε για αυτή τη θέση. Εν ώψη του τριλόγου. Και κατόπιν μπορούμε να θεσπίσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου και να πούμε δεν διαπραγματευόμαστε περαιτέρω για το τι πετύχαμε μέχρι τώρα. Αυτό κάνουμε. Και ελπίζω ότι αν η Επιτροπή ολοκληρώσει τη μελέτη αντικτύπου και δείξει ότι δεν υπάρχει φορολογικός αντίκτυπος, αυτό είναι το φορολογική επίπτωση, ε, δημοσιονομική επίπτωση, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα και μην ξεχνάτε ότι τελικά και αυτό το θέλει ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, διότι ε, έχει ένα εξάμεινο μπροστά του για να γίνει η μελέτη αντικτύπου. Έχουμε και την επιτοπία εδώ, μπορεί να μας πει. Έχω την εντύπωση ωστόσο ότι αν η θέση μας ε, γίνει δεκτή και το Κοινοβού και το Συμβούλιο πάρει την μελέτη, θα μπορεί να δεχθεί τη θέση μας χωρίς άλλη αλλαγή. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να τελειώσουμε σε αυτή τη θητεία το ζήτημα. Περνάει στην επόμενη θητεία αναγκαστικά. Παρότι είχαμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Τυπικά δεν έχουν πει ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε το σημείο αυτό, αλλά ε, στο πίνακα των τεσσάρων στυλών που έχουμε ε, μας είπε ιδίω από το Συμβούλιο κάποιο, ο υπεύθυνο, ότι μπορεί να το δεχθεί το Συμβούλιο. Τυπικά δεν είναι συμφωνία, αλλά δείχνουν ότι μπορούν να δεχθούν αυτό ή εκείνο. Και ελπίζω να δεχθούν και το σύνολο στους 6 μήνες όταν γίνει η μελέτη αντικτύπου. Ας μιλήσουν και οι άλλοι σκιώδεις τότε. Εύλην, οι συμβιβασμοί που πετύχαμε είναι με τους σκιώδεις, σωστά. Δεν είναι... Αυτό αντικατοπτρίζει το που ήμασταν, τι κάναμε, αλλά δεν είναι τι κάναμε με το Συμβούλιο, αλλά μεταξύ μας. Αυτό είναι σαφές, διότι η Εύνη λέει, αν δημιουργήσουμε προηγούμενο, δεν είναι προηγούμενο. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σου, αλλά μην ξεχνάτε ότι μπορούμε να πάμε στην Ολομέλεια και να πούμε κοιτάξτε πόσο κοντά είμαστε και να θούν και να δείξουμε ότι τα κράτη-μέλη είπανε θέλουμε μελέτη αντικτύπου. Αντικατοπτρίζει το που είχαμε φτάσει αλλά στο εσωτερικό μας, όχι έναντι του Συμβουλίου. εν ολίγης. Και συνοπτικά. Σε συνοπτική παρουσίαση. Είναι που, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει. Ήταν, ε, κρίθηκε απαραίτητο να επικεντρωθούμε στα θέματα τα οποία είναι τα πιο σημαντικά για μας και αφήσαμε κάποια, γιατί υπήρχαν βέβαια, πλεονασματικά στοιχεία, περιτά στοιχεία, στην άκρη. Νομίζω ότι χάει τι τις δικές μου τροπολογίες ε, εννοεί και αυτές θέλει να βγάλει, αλλά τέλος πάντων. Καλό είναι πάντα να δείχνουμε ότι υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, παίξαμε το θεατράκι μας, τώρα έχουμε το νομοθετικό κομμάτι. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των σκιωδών. Πιστεύω ωστόσο ότι τα αισθήματα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο ήταν αντίστοιχε με την εξαίρεση του κανονισμού και της οδηγίας. Εκεί είναι το μόνο αμφιλεγόμενο σημείο δεν θα πρέπει να σκεφτούμε ωστόσο να έχουμε μια ε, σκληρή δήλωση στην Ολομέλεια. Δεν μ' αρέσουν τα θεατρινίστικα, αλλά που και που έρχονται οι πράσινοι, ξέρετε, που βγάζουν, ε, φοράνε μάσκες ή, φοράνε, ή βγάζουν ε, αφήσει. Ίσως θα έπρεπε το Κοινοβούλιο συνολικά να δείξει τη διαφωνεί με, το, με τη θέση του Συμβουλίου στο σημείο αυτό και θα βγούμε και στις ειδήσει έτσι. να φορέσουμε, να, φορέσουμε πινακίδες αυτοκινήτων. Δεν θέλω να σας ε, μειώσω τη χαρά, αλλά σε μόνιμη θέση εγώ ήμουν αντίθετος με μία διάσταση της πρότασης. Το ότι οι πινακίδες πρέπει να έχουν ενιαίο μέγεθος, τύπο και χρώμα. Αυτό δεν μ' αρέσει. Και αυτό θα το καταψηφίσει η ομάδα μου. Όχι ότι διαφωνούμε τη διαδικασία, αλλά δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ψηφίζω σήμερα, οπότε θα υποστήριξω τη θέση σου. Περίπου. Λοιπόν. Yeah. I think we've got to be clear about that compromise. Κοιτάξτε, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ε, το θέμα των πινακίδων δεν υπάρχει συμφωνία επ' αυτού και είναι σαφές, διότι αν βλέπαμε πινακίδες αυτοκινήτων με το EU, ούτε κι εγώ θα το δεχόμουν. Συμβιβασμός είναι και δεν περιέχει πινακίδες με το EU. Να το βάλουμε σε αιτιολογική σκέψη. αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη. Τέλος πάντων, ψηφίζουμε ονομαστικά. επικαιροποιημένη πρόταση που θα πάει στην Ολομέλεια ονομαστικά. Και αυτή θα είναι η τελική θέση σε πρώτη ανάγνωση. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορία. 27 υπέρ, 4 κατά. Ωραία, ευχαριστώ. Προχωρούμε στο τελευταίο νομοθετικό κείμενο που ετοιμάζουμε. Η συγγήτρια, η κυρία Κόμη. Και θα γίνει παρουσίαση από την Επιτροπή. Όσοι φεύγετε για, από αυτή τη σημαντική συζήτηση για τα εμπορικά μυστικά, το εμπορικό απόρριτο, σας θυμίζω ότι πρέπει να συναντηθούμε στις 5 ε, παρα 10, λάθος, ε, καθυστέρηση δηλαδή. θα, θα γίνει συνάντηση των συντονιστών μετά από αυτό το θέμα. I just want to see who is going to lead for the commission. Ποιος θα μιλήσει από την Επιτροπή. Η κυρία, ο κύριος Φερνάντες. Fernandez, Salas, is that right? Okay. You're down here as Ms. I'm sorry about that. Σας έχουν ως κυρία εδώ πέρα, συγγνώμη κύριε Φερνάντες. Θα μας πείτε την πρόταση και περί τίνος πρόκειται. Να καλέσω ωστόσο την κυρία Κόμη ω εισηγήτρια από την νομική επιτροπή να μα ενημερώσει. Λίγη ησυχία ρε παιδιά. Για να μας ενημερώσει για το πώς έχει κατάσταση με την νομική επιτροπή. Και τι προτείνεται. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται για να ξεκινήσουμε μπας και κερδίσουμε λίγο το χαμένο χρόνο. Παρότι η προεκλογική εκστρατεία είναι κοντά μας, ε, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για το θέμα αυτό, διότι με εντυπωσίασε το θέμα. Ήξερα ότι στην Ιταλία υπήρχε μια προστασία του εμπορικού απόρριτου και μου φαινόταν περίεργο και, και απεριτώ να έχουμε και άλλη σχετική νομοθεσία. Ωστόσο διαπίστωσα και η διαπίστωση αυτή ήταν ε, δυσάρεστη κατά κάποιο τρόπο ότι δεν σημαίνει το ίδιο σε όλη την Ευρώπη. Η Ιταλία είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που προβλέπει ειδικού κανόνες για, για το εμπορικό απόρριτο. Με εξέπληξε πολύ αυτό και προσπάθησα να καταλάβω το δοσί αυτό. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρόταση χωρίς την οποία δεν θα είχε νόημα να μιλήσουμε για ε, ένωση ένοψη του 2020. Δεν υπάρχει προστασία του, του πνευματικού, των πνευματικών δικαιωμάτων με διαφορετική νομοθεσία στην Ευρώπη. Πλέον η έρευνα και η ανάπτυξη είναι πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομίας και αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε με τον τρόπο αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο ε, και η πρόταση αποδεικνύει ότι έχει ευρύ φάσμα λόγω της χρήσης διατυπώσεων που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες TRIPS. διαβάζοντα την πρόταση φαντάστε καμία από τι πολλέ μικρομεσαίες επιχειρήσει, εξαιρετικά μικρέ ορισμένε περιπτώσει, για τι οποίε ε, η ιδέα είναι βάση τη επιτυχία και προσπάθησα να καταλάβω τι συμβαίνει αν μια ιδέα ε, είναι ιδέα που συγκρούεται με αντίστοιχη άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εσωτερική αγορά. Ε, να μη... Συγγνώμη γιατί μιλάω γρήγορα, το κατάλαβα. Συνεχίζω. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εσωτερική αγορά αν οι κανόνες είναι διαφορετικοί. Ούτε θέλω να φανταστώ τι θα κόστιζε κάτι τέτοιο σε θέμα χρόνου από χρόνο και πόρους όταν ε, χρειάζεται να στραφεί δικαστικά εναντίον του εταίρου αυτού. Επιπλέον, άλλη περίπτωση, μια ιδέα που δεν έχει ακόμα τι τις για να πάρει δίπλωμα και ε, υποκλέπτεται. Δεν μπορεί να μην υπάρχει τέτοια προστασία. Η οδηγία αυτή λοιπόν είναι εξαιρετικά θετικό νομικό εργαλείο, πόσο μάλλον που η προσέγγιση που επιλέγεται δεν είναι, είναι προληπτική και όχι τιμωρητική, ακριβώς για να εξασφαλιστεί ότι η εμπιστοσύνη πρέπει να εντάσσεται στην εσωτερική αγορά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια μικρή λεπτομέρεια και μπαίνω στι λεπτομέρειε τη πρόταση. Μιλώ για την ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του δικαιούχου του απορρίτου αφενό και τη ελευθερία έκφραση και παρουσίαση των πληροφοριών αφετέρου, την προστασία των θεμητών συμφερόντων και την υλοποίηση των μη συμβατικών υποχρεώσεων αφετέρου. Όπω και για κάποια γλωσσικού χαρακτήρα θέματα, ιδίω στην κατάσταση των ε, κοινότοπων ε, πληροφοριών ή του νομικού εκπροσώπου που σε διάφορες γλώσσες μπορεί να έχει διαφορετική έννοια. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι πρέπει να, να ε, περισσότερο την περίοδο περιορισμού των προτάσεων της οδηγίας. Μία υπερβολικά κοντινή ανώτατη προθεσμία μπορεί να μην επιτρέψει ε, επιχειρήσει να μαζέψουν ε, όλο το αποδεκτικό υλικό ενώ μια πολύ απόμακρη ημερομηνία μπορεί να καταστήσει την ε, συζήτηση μάταιη. Πρέπει να αναγνωρίσω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη στο κείμενο και τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του δικαιώματος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, Αυτά που ανέφερα είναι λεπτομέρειες. Εδώ μπροστά μας έχουμε μια πρόταση που επιτρέπει να ανεβεί το, να υψωθεί το επίπεδο προστασίας ε, και αφήνει παράλληλα τα κράτη-μέλη ε, ελεύθερα να εφαρμόσουν ε, να επιβάλλουν υψηλότερους κανόνες προστασίας. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να προχωρήσει γρήγορα στην έγκριση του νομιθού και ευχαριστώ τους συναδέλφους που θα συνεργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή ήδη από τώρα. Να ακούσουμε βέβαια και την Επιτροπή, τους συναδέλφους και θα κλείσω και με μια πρόταση για την ε, Νομική Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα εισαγωγικά. Πρωτού προχωρήσουμε με τη συζήτηση. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Βέβαια έχουμε και μια συνάντηση στις 7 Απριλίου, αλλά η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, που είναι επικεφαλής επιτροπή, θα συντάξει κάποιο κείμενο ή προτείνετε εσείς να στείλουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία στο χρόνο που μας απομένει. Θα ήταν χρήσιμο. Έχουμε κάποιους σκιώδεις μαζί μας εδώ. Ε, μπορείτε να μας πείτε ακριβώς τι προτείνετε εσείς, τι θέλετε από εμάς. Με προλάβατε. Η πρόταση αυτή θα ήταν μια πρόταση που θα έκανα και στο τέλος, ακούγοντα του και ηγητές. Ακριβώς διότι βρισκόμαστε στο τέλος, είναι καλό να υπάρξει μια επιστολή με τις θέσει και τις τάσει μας για την νομική επιτροπή. Και για να επιταχύνουμε το χρόνο, δεδομένου το ότι στι 7 κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσουμε. Είτε σπάντων μπορεί να υπάρχουν άλλα εμπόδια. Ό,τι θέλουν οι ισχυροί βέβαια. Αυτή είναι η πρότασή μου. Επιστολή που πρέπει να στελεί στην νομική επιτροπή όπου λέμε σαφώς τα σημεία που είναι σημαντικά για την ε, εσωτερική αγορά και την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ήθελα να ε, ξέρω ποιος παρακολουθεί, ο κύριος Φόξ παρακολουθεί, ο κύριος Armstrong από τους Πράσινους είναι κανείς που παρακολουθεί το θέμα από τους σοσιαλιστές. Uh, Ο κ. Μάντες βέβαια εκ μέρους των φιλελευθέρων το παρακολουθεί. Ας ακούσουμε λοιπόν από τον κ. Φενάντη Σάλλες από τη Γενική Διεύθυνση ε, αγοράς, τουρκικής αγοράς. Ε, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αλλά περιμένουμε να ακούσουμε την παρουσίασή σας για την πρόταση και μετά ίσως να έχουμε μια, ένα μικρό γύρο συζήτησης. Ε, έχουμε τις διαφάνειες και οι συνάδελφοι έχουν και αντίγραφα των διαφάνειών. Thank you, Mr. Chairman. I'll try to be short. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος και θα επικεντρωθώ στα θέματα από πλευράς εσωτερικής αγοράς. Το, εμπορικό απόρριτο είναι σημαντικό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, πολύ σημαντικό σε διαφορετικά επίπεδα και για την καινοτομία και για την ανταγωνιστικότητα και θέλουμε να τονίσουμε κάτι το οποίο είχε, έχει αναφέρει, ήδη έχει αναφέρει η κυρία Κόμη. την ανάγκη συνεργασίας ε, σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς μεταξύ των επιχειρήσεων. Τώρα, υπάρχει θέμα επεξαίρεσης του εμπορικού απόρριτου υπάρχουν ε, έρευνες που δείχνουν ότι ε, μία στις πέντε επιχειρήσεις πλήττονται από αυτό το πρόβλημα. Ποια είναι η νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Αυτό που παρατηρούμε όταν το μελετάμε εμείς το θέμα ε, για το θέμα της νομικής προστασίας είναι κατακαιρματισμένο και ανεπαρκές σε επίπεδο κρατών μελών. Στα δεξιά έχουμε κάποια περιγραφή των αδυναμιών και έχουμε μια εικόνα που ίσως να μιλάει από μόνη της. Τα λευκά τετράγωνα είναι αυτά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ε, νομοθεσία ε, ε, στο θέμα προστασίας του εμπορικού απορρίτου και το λευκό είναι η απουσία νομοθεσίας. Αυτό επηρεάζει την εσωτερική αγορά. Πιστεύουμε ότι ναι. Πρώτα απ' όλα, τα κίνητρα για καινοτόμες ε, διασυνοριακές ε, δραστηριότητες ε, υποσκάπτονται. Σύμφωνα με τις μελέτες, 40% των επιχειρήσεων δεν μοιράζονται εμπορικά μυστικά για, με άλλους εμπορικούς εταίρους και αυτό οδηγεί σε λιγότερο ενδιαφέρον ε, προς διασυνοριακή συνεργασία. Επηρεάζεται και η ανταγωνιστικότητα. Το, οι νόμοι περί εμπορικού απόρριτου οδηγούν επίσης σε νόμους ε, σχέσεων μεταξύ πολίσεων και ε, πελατών. Ποια, τι προσπαθεί να πετύχει η οδηγία νομική προστασία που θα μπορούσε να συμβάλλει σε βελτίωση των συνθήκων έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ε, τι προτείνουμε. Δεν προτείνουμε την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου. Επικεντρωνόμαστε στην ευαισθητοποίηση για τα θέματα ε, εθνικής νομοθεσίας. Αυτό θα ήταν ανεπαρκές αλλά εναρμόνιση του αστικού δικαίου και της προστασίας του αστικού δικαίου. Έχουμε τη νομική βάση που είναι το άρθρο 114 της Συνθήκης. Τώρα, εν συντομία, τι αναφέρεται στην οδηγία αυτή. Πρώτα απ' όλα, είναι μια συμφωνία TRIPS, ένα κείμενο που συμμορφώνεται με συμφωνία TRIPS, η οδηγία ορίζει το πεδίο εφαρμογή της προστασίας σε τρία επίπεδα. Τι σημαίνει εμπορικό απόρριτο, ορισμός του μη νόμιμου, μη νόμιμη απόκτηση εμπορικών στοιχείων και το θέμα του ασφαλούς λιμένος. Και η κυρία Κόμη ήδη αναφέρθηκε στην ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία πληροφορίας και την ε, μη νόμιμη ε, συμπεριφορά. Υπάρχουν και ένδικα μέσα που προβλέπονται από την οδηγία. Επιπρόσθετα υπάρχουν και άλλες διαδικαστικές ε, ασφαλιστικές δικλείδες που είναι πολύ σημαντικές το τομέα των εμπορικών απορρίτων, όπως για παράδειγμα την διατήρηση της εμπιστευτικότητας ε, των εμπορικών απορρίτων. Τέλος, υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές ε, δικλείδες για να διασφαλιστεί η αναλογικότητα όλης αυτής της δέσμης μέτρων. Ποια είναι τα ωφέλη που αναμένονται από αυτή την οδηγία θα πρέπει να έχει, οδηγήσει σε βελτίωση της νομικής προστασίας του εμπορικού απόρριτου. Υπάρχουν και άλλα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτό, ε, όπως οι γνώμες ε, των κατόχων εμπορικών απορρίτων. Εδώ που εξηγούν ότι αυτό το ασφαλέστερο περιβάλλον θα προκύψει θα βελτιώσει ε, τις ε, διαδικασία των αγωγών σε διασυνοριακό επίπεδο. Υπάρχει καλύτερη διασυνοριακή προστασία των ε, ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων. Και έχετε στη διαφάνεια τα διάφορα ποσοστά. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βελτιωμένης δραστηριότητας στον τομέα της καινοτομίας. Είναι όλοι πεπισμένοι γι' αυτό. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Όχι, δεν έχουν πιστεί όλοι. Οι κάτοχοι εμπορικών απορρίτων, οι επιχειρήσεις γενικά, ε, είναι πεπισμένοι για αυτά που σας έχω και υποστηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα, όταν κάναμε μια δημόσια διαβούλευση στο θέμα αυτό, οι πολίτες που απάντησαν, είχαμε περίπου 150 πολίτες που απάντησαν, δεν ήταν πλήρως σίγουροι και πεπισμένοι για διάφορους λόγους. Αλλά ε, θέλαμε να το υποδείξουμε αυτό σε εσά και από πλευράς επιχειρήσεων υπάρχει στήριξη για αυτή την πρόταση. Αυτά είχα να πω, μια σύντομη παρουσίαση και είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Okay, I think was very clear. Πολύ σαφής. Σας ευχαριστώ και για τις διαφάνειες, διότι ήταν ε, μεστές ε, στοιχείων. Ποιος θα ήθελε να συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση, ποιος θα ήθελε να προσθέσει, να πει την άποψή του, κύριος Έμστρον, κύριος Σβάπ, κύριος Φόξ, Μάντας. Κάποιος άλλος. Ευχαριστώ. Και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Κόμη. Κυρία Έγκστρομ. Ε, Πολλά πράγματα μπορεί να πει κανείς επί της ουσίας. Δεν είναι απαραίτητα καλή ιδέα να μπει μια γενική ρύθμιση για τα ε, δικαιώματα πνευματικής διοκτησίας. υπάρχουν η βιομηχανική διοκτησία, υπάρχει το ένα το άλλο. Ε, το σήμα δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα άλλο, γιατί δεν είναι ότι προσπαθούμε κάτι να κρύψουμε εκεί μέσα. Υπάρχουν πολλές συνέπειες που αφορούν ακόμη και τους εργαζομένους όταν θα θέλουν να αλλάξουν δουλειά, θέσεις εργασία. Μια μεγάλη πρόταση λοιπόν με πολλές συνέπειες. Και για να μην ειλικρινής, μου φαίνεται ότι κατατίθεται σε πολύ όψιμο χρόνο. Δεν έχει λόγο το κοινοβούλιο να τοποθετηθεί, ούτε καν χρωμοδότηση δεν χρειάζεται να κάνουμε, γιατί όποια χρωμοδότηση και να εκφράσουμε εμεί. δεν ε, υπάρχει εγγύηση ότι θα συμφωνήσει το προσεχέ κοινοβούλιο. Νομίζω ότι χάσιμο χρόνο θα είναι να εκφράσουμε εκ μέρου του κοινοβουλίου στην παρούσα θητεία γνώμη. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να τα αφήσουμε για την επόμενη. Κύριο Σφάπ, ευχαριστώ πρόεδρε. με μου φαίνεται ήταν πολύ ενδιαφέρον και διαφωτιστικό το έργο της κυρίας Κόμη τόσο μας παρουσίασε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η ενοποίηση της, ε, του δικαιικού πλαισίου στο κράτη-μέλη και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ε, επαγγελματικό μυστικό έχει λόγο ύπαρξης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ταυτόχρονα είναι μια καλή και ισορροπημένη πρόταση σε κάποια σημεία ίσως θα πρέπει να κάνουμε μικρορυθμίσεις. Η κυρία Κόμη έχει επεξεργαστεί κάποια σημεία, χρειάζεται να είναι πιο σαφείς κάποιοι ορισμοί, όχι υπερβολικά ευρύς. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε μια πολύ αφηρημένη νομική περιγραφή του τι είναι μια μερικές φορές παγιωμένη επαγγελματική πρακτική. Και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει από νομικής να ολοκληρώνουν στη δικασία επιχειρήσει προκειμένου να αποδεικνύουν ότι υπήρξε κλοπή ε, ε, η υπεξαίρεση ε, επιχειρηματικών μυστικών. Αυτά και εδώ νομίζω ότι πολύ σωστά επισήμανε και ο κ. Σέγκστρομ ότι η οδηγία δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τον, εργαζόμενο να αλλάζει ε, θέση εργασίας ε, εφόσον έχουν αναλάβει κάποιο ερευνητικό έργο κτλ. Και θα πρέπει και η επιχείρηση να αποδεικνύει ότι υπάρξει μία παράτυπη, παράνομη αφαίρεση επιχειρηματικών μυστικών. Άρα πλήρες βάρος αποδείξεως θα πρέπει, το πλήρες βάρος αποδείξεως θα πρέπει να το φέρει η ίδια η επιχείρηση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Δεύτερον, σε ποιο βαθμό και, σε ποιες προϋποθέσεις, και με ποιες προϋποθέσεις επαγγελματικά μυστικά τα οποία ε, μπορεί να παρεμποδίσουν ή να ελέγξουν την περαιτέρω εξέλιξη αποκλείονται ή αφαιρούνται. Δηλαδή, το λεγόμενο new economy και το old economy. Δηλαδή, ξέρω πώς μπορώ να γράψω ένα σύστημα μέσα σε, ένα μηχάνημα, να δώσω οδηγίες λαμβάνω τις σχετικές οδηγίες από την αρμόδια επιχείρηση με τη βεβαίωση ότι δεν τίθενται τα στοιχεία αυτά και σε άλλους, ότι είναι δηλαδή μυστικά απόρριτα, αλλά εάν τυχόν με παράλληλη ε, έρευνα κάποιος άλλος εξασφαλίσει το ίδιο know-how, την ίδια τεχνογνωσία, τότε θα πρέπει να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε τις ε, διαφορές. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε εάν κανόνες που ήδη υφίστανται στα κράτη-μέλη, γιατί υπάρχουν παντού, απλώς διαφοροποιούνται κατά περίπτωση, μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να αποφύγουμε περιστάσεις όπου στη Βουλγαρία, και δεν θέλω να υψηλθώ λεπτομέρειες, αλλά το δίνω μόνο σαν παράδειγμα, μια κινέζικη επιχείρηση αποδεικνύοντας με, με αποδεδειγμένα κλεμμένα κλεμμένη τεχνογνωσία από γαλλική επιχείρηση μπόρεσε να εξασφαλίσει ακόμη και ευρωπαϊκή επιδότηση για την κατασκευή ενός αποτεφρωτήρα αποβλήτων στην Βουλγαρία και δεν ήταν σε θέση οι βουλγαρικές αρχές να συνδέσουν την κλοπή αυτή της τεχνογνωσίας των επαγγελματικών μυστικών με την αφαίρεση της άδεια και της ενίσχυσης. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει εν τέλει καινοτομία ανταγωνιστών που αποτελεί αντικείμενο κλοπής δεν πρέπει να αξιοποιείται εις βάρος αυτών που την έχουν φτιάξει. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μία λύση ώστε να μην καίγονται μαζί με τα ξερά και τα χλωρά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Μαζί με το ΕΛΚ πιστεύω ότι θα πρέπει να αποστείλουμε την επιστολή στην καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή. Όπως είπε ο κύριος Έγκστρεμ πολύ σωστά δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε με την γνωμοδότησή μας την προσεχή σύνθεση του Κοινοβουλίου, αλλά ταυτόχρονα δεν νομίζω ότι θα πρέπει και να σιωπήσουμε. Να σιωπήσουμε. Πρέπει να εκφράσουμε τις θέσεις μας, να αποστείλουμε την επιστολή και να συστήσουμε στο βαθμό που μπορούμε, γιατί αποτελεί μια πρόταση λογική, άλλωστε σχετική με τα όσα μας είπε ο Έντμου Στόιμπερ σήμερα, δηλαδή το να αποφεύγουμε την υπερβολική γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Fox. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ. Η ομάδα μου υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής και υποστηρίζω αυτά που είπε ο κ. Φάμπερ, να στείλουμε μια επιστολή με την υποστήριξή μας, χωρίς να δημιουργήσουμε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των εμπορικών, του εμπορικού απορρίτου σε όλα τα κράτη-μέλη. Όπως είπε η Επιτροπή, κάτι τέτοιο βοηθά την ανάπτυξη. Μια λέξη μόνο, προσοχή κάποιος συνάδελφος μίλησε για εμπορικό μυστικό στην ίδια πρόταση με την ε, πνευματική και διανοητική διοκτησία. Διαφορετικά πράγματα. Δεν πρόκειται για πνευματική ιδιοκτησία. Αυτές είναι δημόσια καταγεγραμμένες και πρέπει να ορίσεις από τι προστατεύεσαι. Το επαγγελματικό μυστικό είναι εξορισμού μυστικό δεν είναι δημόσιο. Μπορεί να είναι ε, τα συστατικά μιας μπάρα σοκολάτας ή ένας, αυτό χρειάζεται διαφορετικό τρόπο προστασίας και δεν πρέπει να μπερδεύουμε πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικό μυστικό. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Κύριε Βερνιό. Θα είμαι πολύ σύντομη, Πρόεδρε. Η πρόταση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η συζήτηση που είχαμε είναι γεγονό ότι δείχνει πως πρέπει να διευκρινίσουμε πολλά πράγματα. Ορισμούς κατά βάση. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Έγκστρομ. Δεν μπορούμε ένα μήνα πλην λήξη θητεία να μπούμε σε ένα τέτοιο φάκελο που θα μας οδηγήσει σε αξιολογήσεις, σκέψεις και παρατηρήσεις εξαιρετικά εκτεταμένες. Θα πρέπει να αφήσουμε στην επόμενη Επιτροπή ΙΜΚΟ απόλυτη ελευθερία για να συζητήσει, όχι βεβαιασμένα, σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με την θέση του κ. Έγκστρομ. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Να τα αφήσουμε στην επόμενη επιτροπή για να δει ε, με ηρεμία ορισμούς, διευκρινήσεις και να έχει ένα κανονικό σωστό διάλογο. Ο κύριος Μάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνταγή της coca είναι εμπορικό μυστικό. Τώρα, το ότι έχει πολύ ζάχαρη μέσα, αυτό δεν είναι απόρριτο και μυστικό. Αυτή είναι μια δήλωση, αλλά αυτό που θέλω να προσθέσω, γιατί ασχολούμαστε αρκετά χρόνια με αυτό το θέμα, είναι αξιόλογο θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να έχουμε κόσμο εδώ στην Επιτροπή, διότι όλοι συμμετέχουν στην προεκλογική εκστρατεία. Σε 8 εβδομάδες έχουμε εκλογές. Ίσως να γράψουμε μια επιστολή που να είναι σημαντική και να την διατηρήσουμε. Αυτό το στηρίζω κι εγώ. Αλλά μια έκθεση αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο, μας πιέζει ο χρόνος, δεν είμαι υπέρ της για την σύνταξη μιας επιστολής που θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα και θα μπορούσε να παραμείνει σε αυτή την Επιτροπή και συμφωνώ με τον Άσχλη, δεν είναι θέμα ε, δικαιώματος διανοητικής ε, ιδιοκτησίας, είναι εμπορικό απόρριτο και θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό μέσα στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Αλλά τώρα να έχουμε ολόκληρη έκθεση με και συζητήσεις, δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό. Η άποψή μου. Okay, well, I think Θέλει κανείς άλλος να παρέμβει. Νομίζω θα συμφωνούσαμε με τους συναδέλφους ότι δεν θα μπορούσαμε να το δούμε εις βάθος το θέμα. Μου φαίνεται το θέμα για την επικεφαλής ε, επιτροπή δεν θα αλλάξει στην επόμενη θητεία, γιατί έχουν ήδη οριστεί οι υπεύθυνε αρμόδιες επιτροπές. Το πραγματικό θέμα, και θα ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Κόμη, σε αυτό δεν έχει νόημα εδώ να γράψουμε μονομερώς μια επιστολή αφού δεν είμαστε η επικεφαλής επιτροπή. Τώρα, εάν η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα ε, προτείνει κάτι, τότε θα παραμείνει στο φάκελο για την επόμενη επιτροπή να το παρακολουθήσει. Αν το κάνουν αυτό, τουλάχιστον θα φαίνεται ότι έχουν συνεισφέρει σε αυτό, διότι εμεί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι συμφωνούμε και ακολουθούμε πλήρως το φάκελο στην επόμενη θητεία. Και σχετικά με το ε, αν σας αρέσει είτε όχι. Βέβαια πάντα μπορείτε να προσθέσετε τις επιφυλάξεις σας ε, και ήθελα η κυρία Κόμη να μας διευκρινίσει ακριβώς ποια είναι η πρόθεση του εισηγήτη ή του οριστέντος δι, ε, εισηγητή στην Επικεφαλής Επιτροπή, έτσι ώστε να ξέρουμε πώς να ανταποκριθούμε. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό θα είναι χρήσιμο και οποιαδήποτε άλλα σημεία θέλετε να μας προσθέσετε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Σύμφωνα απόλυτα ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε συζητήσεις και τροπολογίες ε, χωρίς να έχουμε χρόνο. Θυμίζω ωστόσο ότι είμαστε βουλευτές μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δουλειά μας μεταξύ άλλων είναι να φτάσουμε στο τέλος της θητείας μας με ενδείξεις που θα μπορούσαμε να δώσουμε ως προς το single market και αυτό που έγινε στην θητεία μας. Διότι τα κείμενα που εγκρίναμε και από τον Επίτροπο Μπαρνιά και από τον Μάριο Μόντι οδήγησαν σε αλλαγέ στην θητεία. Και δεύτερον θα πρέπει να δώσουμε και γενικές κατευθύνσεις. Αυτό δεν είναι χαμένη δουλειά, αλλά και μια κληρονομιά που μπορεί να αφήσουμε στην αρμόδια επιτροπή. Αλλά δημοκρατία έχουμε, η πλειοψηφία αποφασίζει ό,τι θέλετε. Um, δεν απαντήσετε στη βασική μου παρατήρηση. Η γραμματεία μου λέει ωστόσο ότι οι νομικοί, οι συντονιστέ τη νομική επιτροπή συζητούν αυτό αύριο. Η δική μου σύσταση ως πρόεδρο είναι, αν συμφωνείτε, να περιμένουμε την απόφασή τους αν αποφασίσω να ετοιμάσω ένα κείμενο εργασία και οτιδήποτε είδους μπορείτε να πείτε ότι δεν θα γίνει αυτό από πλευρά μας και να μας πείτε και το χρονοδιάγραμμα. Και αν δούμε το κείμενο εργασία να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Αν δεν υπάρξει κείμενο εργασία θα συμφωνήσουμε με τους συναδέλφους που λένε ότι δεν θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε κάτι από μόνοι μας γιατί δεν έχουμε το χρόνο. Αυτό νομίζω είναι η σωστή προσέγγιση. Δεν ξέρω αν το θέλουν, θέλουν να το συζητήσουν χωριστά οι συντονιστές αυτό. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγώ συμφωνώ πρόεδρε. Δεν είχα καταλάβει ότι οι συντονιστές της νομικής συναντιούνται αύριο εφόσον αυτό γίνει έχουμε χρόνο να αποφασίσουμε έγκαιρα. Αν γινόταν αυτό την άλλη εβδομάδα δεν θα είχαμε χρόνο. Σύμφωνα λοιπόν με την πρότασή σας που νομίζω ότι είναι και πιο εφικτή. Ωραία, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την Επιτροπή και του συναδέλφους που ήθελαν να μα μιλήσουν για το θέμα αυτό. Έχετε τα κείμενα, περιμένουμε τι θα πει η νομική επιτροπή αύριο. Κλείνουμε για σήμερα. Συντονιστές. Είναι εδώ όλοι οι συντονιστές νομίζω. Σας θυμίζω ότι η επόμενη και τελευταία συνάντηση της Επιτροπής μας είναι Δευτέρα 7 Απριλίου στις 3 το απόγευμα. Και θα έχουμε και μια μικρή δεξίωση μετά εδώ απ' έξω, έξω από την αίθουσα της Επιτροπής. Και θα έρθουν τρεις Επίτροποι να μας πούν τις ιδέες τους. Και να σκεφτούμε τι κάναμε. Η μέτα, Σεμέτα, Μίμητσα και Μπαρνιέ. Όλοι τους. Και ο κύριος Μίμητσα θα μας μιλήσει και για το βαθμολόγιο για την προστασία των καταναλωτών οι συντονιστές καλό θα ήταν να τραβήξουν και μερικούς βουλευτές να μην, να είναι, μην είμαστε αρέα αρέα. Ε, πείτε τους και για τη δεξίωση. Θα έχουμε και κάποιες φωτογραφίες ε, από την κοινή δουλειά μας και θα μιλήσω και εγώ να σας πω τι κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Προφανώς είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσετε. Θα τα πούμε τον Απρίλιο Λύεται η συνεδρίαση και σε λίγο ξεκινάμε τους συντονιστές.